Okay, good morning everybody. Λοιπόν, καλημέρα συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Κρίμα που έχουμε πολύ λίγους συναδέλφους εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σε κάθε περίπτωση. Πρώτον, να ζητήσω συγγνώμη εξ της, της κυρίας Πακ που δεν μπορεί να προεδρεύσει σήμερα στην συνεδρίαση, θα είναι εδώ το απόγευμα. Ε, μία σημαντική αλλαγή στην ημερησία διάταξη Δυστυχώ, ένας από τους υπουργούς του, της Προεδρία Προεδρίας του Συμβουλίου με τον οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε απόψε ο κ. Κουίν δεν θα μπορέσει να είναι παρόν για οικογενειακούς λόγους. Θα τον αντικαταστήσει ο υφυπουργό, κύριος Κένεν, υφυπουργό ε, κατάρτισης και δεξιοτήτων. Με αυτή την αλλαγή Μπορούμε να εγκρίνουμε την υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Δεν βλέπω να είναι κανείς αντίθετος. Κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής της 26 και 27 Νοεμβρίου του 2012. Προτείνω, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στη συνάντηση, να κριθούν ότι εγκρίθηκαν μέχρι τέλους συνεδρίασης σε ό,τι αφορά την διερμηνία. Σήμερα έχουμε περιορισμένη διερμηνία. Δεν έχουμε διερμηνία για τα βουλγαρικά, τσέχικα, λιθουανικά, λετονικά, μαλτέζικα, σλοβενικά και σουηδικά. Έχουμε. Δεν έχουμε πορτογαλικά το απόγευμα και δεν έχουμε σλοβάκικα το πρωί. Αυτή είναι η γλωσσή, το γλωσσικό μας καθεστώς. Ξεκινούμε. Κάτι άλλο. Είναι το θέμα της σειράς των ε, Μπαίνουμε στο σημείο 4 τη σημερινή διάταξη. διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά. Η συγκριτή είναι ο κύριο Μπέλετ για ανταλλαγή απόψεων. Όπω ξέρετε, ε, το online, ε, τα τυχερά παιχνίδια online είναι βασικό ζήτημα, κυκλοφορεί πάρα πολύ και η βασική προσέγγιση δεν, ε, στην εσωτερική αγορά δεν είναι πλήρω ικανοποιητική. Η ανακοίνωση τη επιτροπή. θέτει μια, ε, ένα πρόγραμμα δράση για τη διευκρίνηση της ρύθμιση ε, του διαδικτυακού τυχερού παιχνιδιού και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή μα ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, είμαστε υπεύθυνοι για θέματα νεότητας. Το 75% των Ευρωπαίων κάτω των 17 χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Μερικοί από αυτούς ε, διατέχουν τον κίνδυνο να κολλήσουν στο παιχνίδι. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ε, δημιουργία καλύτερων ε, εργαλείων παρεμπόδισης και είναι υπεύθυνη για την, έγινε αρμόδια για την υπεύθυνη διαφήμιση και για την ενημερώση για τους κινδύνους της, ε, των τυχερών παιχνιδιών. Εμείς υποστηρίζουμε την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και επί την ανακοίνωση περιλαμβάνει τρόπους για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με μηχανισμούς για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η υπεύθυνη επιτροπή είναι η Γιούρη. Εμεί ετοιμάζουμε μία μη, μία μη νομοθετική γνωμοδότηση με εισηγητή τον κύριο Μπέλετ, όπω σα είπα, ο οποίο θα παρουσιάσει τι αρχικέ του σκέψει. Σήμερα θα παρουσιάσει ένα σχέδιο γνωμοδότηση το Μάρτιο και θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Ήβο, έχει το λόγο. Thanks, uh, very much, very much, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιρετική εισαγωγή σας, έτσι ώστε να μπούμε πια σε λεπτομέρειες. Νόμιζα ότι η καθήλυνα αρμόδια ήταν η ΙΜΚΟ, γιατί έχουμε και μια κοινή γνωμοδότηση με την ΕΚΟΝ. Εντάξει, ωραία. Σωστά τα, τα ξέρω. Λοιπόν, όπως είπατε, Πρόεδρε, και θα είμαι και όσο πιο ακριβής γίνεται, δύο βασικές ανησυχίες υπάρχουν, ο αθλητισμός και η προστασία των ενηλίκων. Σε αυτά τα δύο θα ήθελα να επικεντρωθώ τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνουν πολλού κινδύνου για του ανηλίκους και από τα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια γιατί το όριο για την, για την ένταξή του και για να μπορούν να παίξουν στο ίντερνετ είναι πολύ πιο χαμηλό. Μπορεί δηλαδή κανεί να παίξει και τυχερά παιχνίδια ακόμα και από το τηλέφωνό του. Είναι λοιπόν πολύ πιο απλή η πρόσβαση για του ανηλίκους. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να εφαρμόσουμε σε αυστηρούς ελέγχους ε, για την ε, ηλικία και για την ταυτότητα ε, μέσω ας πούμε ενός ηλεκτρονικού σήματος. Αυτό σε κάποια κράτη μέλη υπάρχει, σε κάποια όχι. Υπάρχει λοιπόν μια αρκετά διαφοροποιημένη προσέγγιση σε όλο το επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτό. Και να προσθέσω επίσης ότι η εκπαίδευση πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο όταν μιλούμε για την πρόληψη που θα πρέπει βεβαίως να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε που σχετίζονται με τον τζόγο. Οι ανήλικοι πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ειδικά για τα, για τα sites που, είναι, που δεν είναι ρυθμισμένα στην, και είναι στη μαύρη αγορά. Ε, γιατί αυτό βεβαίω δεν έχει να κάνει μόνο με του ανηλίκου, έχει να κάνει με όλου όσου ασχολούνται με θέματα διαδικτυακού τζόγου. Υπάρχει και το θέμα του εθισμού. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε κάποια μέτρα ώστε να αποτρέψουμε ανθρώπους από το να χάνουν τα χρήματά τους. Περίπου 2% και είναι πολύ το 2%. 2% του πληθυσμού της Ένωσης έχει ε, προβληματική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα στοιχήματα. Γιατί και αυτό δεν επηρεάζει μόνο το άτομο αυτό, αλλά και την οικογένειά του βεβαίω και του ανηλίκου ε, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, ανώφλια για το πόσα μπορεί κανείς να βάλει στον λογαριασμό του σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να παίξει. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στα πλαίσια και της, των ε, ημερήσιων όριων που δεν θα πρέπει να μπορεί κανείς να ξεπερνά. Θα πρέπει δηλαδή να μπει ένα ανώτατο όριο που να μπορεί κανείς να τζογάρει στο ίντερνετ. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες τις ε, παρομοίου περιεχομένου στο σελίδες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια, μια κοινή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον κλάδο, μαζί με τις οργανώσεις των καταναλωτών, θα πρέπει να εκφωνήσουν κοινά ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό του εθισμού στον τζόγο. Αυτά λοιπόν είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας ανησυχούν, η προστασία των ανηλίκων και η προστασία γενικώ του πληθυσμού απέναντι στον εθισμό στον τζόγο. Και όπως ε, είπα, η άλλη μας ανησυχία είναι ο αθλητισμός, όπως αναφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε. Ε, ο, οι διαγωνισμοί, οι αθλητικοί διαγωνισμοί είναι ένα από τα βασικά θέματα του, των στοιχημάτων και του τζόγου στο διαδίκτυο. Ε, αποδίδει πολλά έσοδα ε, κάθε χρόνο σε αυτούς που έχουν τέτοιες ιστοσελίδες. Βεβαίως ε, ένα περιορισμένο ε, ποσό των ε, ποσών που τζογάρονται στον στους αθλητικούς διαγωνισμούς, πηγαίνει πίσω, γυρίζει πίσω στους ε, αθλητικές, στις αθλητικές ενώσεις. Οπότε θα πρέπει να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό για το κέρδος που υπάρχει σε ε, επίπεδο διαδικτύου κυρίως για να επιστρέφει σε πολύ βασικές α, ε, μικρές ομάδες ώστε να μην, υπάρχει, ε, να μην μπορεί να υποφεληθούν μόνο οι μεγάλοι όμιλοι από αυτό, αλλά και οι πιο μικρές ομάδες. Και επίσης πρέπει να, πούμε και ε, να μιλήσουμε και για το θέμα των ε, δικαιωμάτων για την οργάνωση τέτοιου είδους διαγωνισμών. Βεβαίω ο τζόγο και τα στοιχήματα μπορεί να έχουν πολύ αρνητικέ επιπτώσει. Ο Μισελ Πλατινί, ο πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ, είπε ότι, ότι ε, συνήθω τα στοιχήματα αυτά είναι στημένα, οπότε προφανώ οι αρνητικέ συνέπειε είναι μεγάλε και ίσω θα πρέπει να υπάρξει κοινή δράση αστυνομικών και δικαστικών δυνάμεων ή και των, αρχών, των εθνικών αρχών, ε, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι εγκληματίες από το να δρουν διασυνοριακά και να καταχρώνται των αθλητικών διαγωνισμών ώστε να ε, ξεπλένουν τα χρήματα, τα που βγάζουν από τον παράνομο τζόγο. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε, μια ευρωπαϊκή, σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα συμπεριλαμβάνει και τα κρατημέλη και την Κομισιόν, από κοινού με την Eurojust, την Europol και με την Interpol. Και προτείνουμε επίσης η απάτη ό,τι αφορά τα, τα στοιχήματα θα πρέπει να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος ώστε αποτελεσματικά πια να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη απειλή για τον αθλητισμό. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Ειδική Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα ε, ε, εγώ είμαι μέλος και σε αυτή την επιτροπή. Το έχουμε λοιπόν και στην δική μας ημερήσια διάταξη εκεί. Και κλείνοντας, Πρόεδρε, να πω κάτι για την πρόταση της Κομισιόν για το σχέδιο δράσης. Η Κομισιόν προτείνει να ανοίξουν οι αγορές και να υπάρξει πρόσβαση σε εμπορικές εταιρείε, όπως και σε, ε, ε, πέραν των δημοσίων δηλαδή που πολλές φορές έχουν ε, το μονοπόλιο σε πολλά κράτη-μέλη και το άνοιγμα αυτό της αγοράς ίσως να είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα, εκτός βεβαίως εάν αποκτήσουμε ένα σταθερό ε, πλαίσιο ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το, αυτή τη μεγάλη απειλή και του διοθισμού στο τζόγο, που είναι απειλή και για τους ανήλικους, αλλά και της, του ξεπλήματος ε, χρήματος. Το τελευταίο, το πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό ήταν η έκθεση Κρόιτσμαν. Και εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οδηγία, δηλαδή μια νομική πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει ελάχιστα πρότυπα που θα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις, όλους τους, παρόχους, τους ρυθμισμένους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών online. Και βεβαίως ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση αυτή. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά θέματά μας για τη δική μας την Επιτροπή τουλάχιστον και βεβαίως ευχαριστώ να ακούσω και τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιβο. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τάκουλα πρώτος. <clears throat> Ε, ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Ιβο για την πολύ σαφή παρουσίασή σου. Είναι μια μοναδική υπηρεσία αυτά τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Μια μοναδική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Καλό είναι να την ελέγχουμε. Πρέπει να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία επί τη βάση αυτής της εκθέσεως. Εγώ ήμουν εισηγητής για μία παρόμοια έκθεση. Νομίζω ότι είναι πολλές ε, οι καλές ιδέες στην έκθεση. Ωστόσο, νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, τους οποίους πρέπει να διορθώσουμε σε μεγάλο βαθμό, σε μεγαλύτερο από ό,τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά. Πρέπει να δούμε τους παράγοντες γύρω από το θέμα αυτό και το θέμα επίσης ε, της ενδεχόμενης καταχώρησης ε, των ε, ανθρώπων που παίζουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε πολλές χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία ιδέα για το ποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές. Και θα έχουμε κάποια ιδέα και για τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τα τυχερά παιχνίδια. και για τον αθλητισμό είναι σημαντικό θέμα. Πολλές μεγάλες εταιρείες ε, συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και συχνά είναι καταχωρημένες ε, με διαφορετικές ονομασίες σε διάφορες χώρες. Ένα παράδειγμα να σας πω. Στη δική μου χώρα. Προσπαθήσαμε να έχουμε πολύ λεπτομερή μητρώα Μπορώ όμω εγώ να είμαι σε ένα μητρό ως ε, Hans Τάκουλα, ως H Τάκουλα ή σκέτο Τάκουλα. Που σημαίνει ότι είναι μάλλον δύσκολο να ξέρει κανείς ακριβώ ποιος συμμετέχει. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ προσεκτικά πώς θα οργανώσουμε αυτή το, αυτό το σύστημα καταχώρησης που πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικό. καταφέρουμε, σίγουρα μπορούμε να μειώσουμε τα εγκλήματα στις, ε, ε, στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής και νομίζω ότι είναι πολύ καλή αφετηρία η έκθεση του Ήβο. Ελπίζω να συνεχίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με, τις, ε, με τη δική μου συνεισφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Ήβο για την παρουσίαση που έκανε με τις βασικές ιδέες της έκθεσής του. Είμαι ο εισηγητής για την, την έκθεση της νομικής επιτροπής και πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κλάδος των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών είναι αυτός με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Υπολογίζεται ότι, ορισμένες, ε, ότι μπορεί να φτάσει και το 40% αύξηση το χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, γύρω στα 7 εκατομμύρια άτομα το χρόνο παίζουν τυχερά παιχνίδια διαδικτυακά. Με, μια, με ένα τζίρο 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για πολλά λεφτά έναν, και είναι ένας τομέας εξαιρετικά ευαίσθητος. Οι χρήστες των, των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών είναι συχνά νέοι, συχνά εθισμένοι, άρα χρειαζόμαστε καλή και ορατή νομοθεσία. Η Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι το 80% των site τυχερών παιχνιδιών δεν έχουν, δεν έχουν έδρα ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι ότι συχνά δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος της Ένωσης στα site αυτά, ενώ παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες της Ένωσης χωρίς έλεγχο και χωρίς φορολογία. Άρα χρειαζόμαστε σωστή νομοθεσία σχετικά. Ε, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε να πετύχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά, πόσο μάλλον να εξετάσουμε υπεράκτια την κατάσταση. Στη Γερμανία, όπου τέτοια παιχνίδια απαγορεύονται, ή σε χώρες όπου τα τυχερά παιχνίδια είναι κρατικό μονοπόλιο, έχουμε άλλες χώρες όπου τα site τυχερών παιχνιδιών είναι μεν νόμιμα και ρυθμιζόμενα και επιτρέπονται ε, ε, ιστοσελίδες με ειδική άδεια, ειδική φορολογία ε, και βασικά κανονικούς ελέγχους. Αυτό είναι νομίζω η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε γιατί αλλιώς, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να ελέξεις ποιος έχει τις άδειες να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την χρήση, για το ποιος χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες αυτές, να υπάρχει νομική παρακολούθηση, να υπάρχει παρακολούθηση των εφισμένων παικτών και τις ηλικίε τους. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι όταν σε μια χώρα τα τυχερά παιχνίδια δεν επιτρέπονται, υπάρχει δυνατότητα κάποιου να χρησιμοποιήσει site που είναι από άλλη χώρα. Άρα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρξει ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν υπάρχουν χώρες που θέλουν να νομοθετούν, ε, που έχουν δική τους νομοθεσία, θα πρέπει να παράσχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των νέων, των ανηλίκων και να υπάρξει επαρκής ενημέρωση για τους κινδύνους του εθισμού. Τονίζω ότι ο τομέας αυτός εξετάζει, εξελίσσεται τόσο δυναμικά που θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι ήδη δίνουμε. Κάτι άλλο. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση του Ήβο. Έχουμε ένα αντίστοιχο, σύστημα στην Πολωνία. Τα χρήματα από τα τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, τα χρήματα, τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια δηλαδή χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση τοπικών δραστηριοτήτων με έμφαση στους νέους. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Κάτι ακόμα. τα αποτελέσματα των αγαθλητικών εκδηλωτιαστηριοτήτων και η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, κάτι που είναι εξαιρετικά διαδεδομένο και το επικίνδυνο. Μήπως θα μπορούσαν να υπάρχουν αντίστοιχες ή παρόμοιες μορφές κυρώσεων σε όλες τις χώρες για αντίστοιχα δικήματα. Για τους αθλητές, για παράδειγμα, που εμπλέκονται σε τέτοιες προσπάθειες ε, στισίματος παιχνιδιών. Και ξέρετε ότι πολύ συχνά χρησιμοποιείται το σύστημα, τα, χρησιμοποιούνται τα στοιχήματα για να αποκομίσουν κέρδη από στήσιμο παιχνιδιών. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην UEFA δομές οι οποίες εξετάζουν το προφίλ διαφόρων στοιχημάτων σε παιχνίδια και μπλοκάρουν τα στοιχήματα όταν βλέπουν ότι υπάρχει ισχυρό κίνδυνος να έχει στηθεί ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Και σε αυτό ε, συμμετέχει, σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει και η Interpol. Όταν υπάρχει λοιπόν υποψία ότι χρησιμοποιούνται παράνομα χρήματα στον αθλητισμό, υπάρχει δυνατότητα να μπλοκάρουμε τα συγκεκριμένα στοιχήματα. Χρειάστηκαν, ε, χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει, δεν, δεν, δεν, δεν λειτουργήσε νόμιμα. Προφανώς ε, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα στοιχήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πλήρη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και η Επιτροπή πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε επαρκώς καλά το σύστημα ώστε να εξασφαλίσουμε σωστό αθλητισμό, προστασία των νέων και προστασία του κλάδου από τα βρώμικα χρήματα του οργανωμένου εγκλήματος και των μαφιών. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το διαδικτυακό τυχερό παιχνίδι θα λειτουργεί με τρόπο που θα προστατεύει τους καταναλωτές, τους χρήστες, τους νέους χρήστες και θα προστατεύει τον αθλητισμό από αυτή την ανώσια συμμαχία με το οργανωμένο έγκλημα. Πολύ σημαντική γνωμοδότηση αυτή του Ήβο. Χρειάζεται να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Συνάλοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, μπορώ να μιλήσω τσεχικά σήμερα, ούτε σλοβακικά, οπότε θα προσπαθήσω στα αγγλικά. Για την ε, ομάδα των ε, σοσιαλιστών θα ήθελα να πω δύο πράγματα. το θέμα αυτό βεβαίως έχει συζητηθεί πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές. Δύο πράγματα όμως θα ήθελα να πω. Συζητούμε την ανακοίνωση της Κομισιόν η οποία λέει ότι το κλάδος αυτός ε, ε, μεγαλώνει, αυξάνεται συνέχεια και από το 2011 στο 2015 περιμένουμε μια αύξηση του 40% σύμφωνα με τούτη την ανακοίνωση. 6,84 εκατομμύρια πολιτών ασχολούνται, παίζουν ε, τζόγο στο διαδίκτυο. Βεβαίω τα κρατημέρια δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό μεμονωμένα. Πρέπει να υπάρξει κοινή δράση, όπως ας πούμε η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου που επηρεάζει και τους ανήλικους αλλά και τους ενήλικους και μέσω αυτού υπάρχει και ξέπλυμα χρήματος κτλ. Σε ένα βαθμό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, η οποία όμως δεν είναι, είναι, μια, είναι προαπαιτούμενο, δεν είναι απλώς θέμα θέλησης. Η Κομισιόν στην ανακοίνωση της λέει ότι τα φαινόμενα αυτά διαδικτυακού τζόγου θα πρέπει βεβαίως να τα δούμε και στα πλαίσια της δικής μας ε, επιτροπής. Πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, τους, ε, τα ανήλικα παιδιά και αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, δεδομένου και του ότι 75% των νέων και των ανηλίκων στην Ευρώπη κάτω των 17 ετών δηλαδή, χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν ότι θα προστατευτούν από οποιαδήποτε ε, κακή πύροη μπορεί να έχει ο διαδικτυακός τζόγος σε αυτά τα παιδιά. Σίγουρα λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιε από αυτέ τι ε, συστάσει για να προχωρήσουμε. Συμφωνώ επίση με την Κομισιόν ότι οι διαφημίσει θα πρέπει να ε, είναι τέτοιε έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και να τους δείξουμε ότι αν δεν παίξουμε υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο τότε όντω ε, η επιρροή μπορεί να είναι πάρα πολύ ε, κακή. Και αυτό πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο θέμα που ήδη αναφέρθηκε είναι η διατήρηση της αξιοπρέπειας του κλάδου του αθλητισμού. Έγινε μια δημόσια ακρόαση για, την, για το fair play και για τον αθλητισμό όπου έκαναν κάποιες προτάσεις οι εμπειρογνώμονε για την αντιμετώπιση των αστημένων παιχνιδιών και του παράνομου στοιχήματο και του παράνομου τζόγου. Ε, αυτή η προβληματική τομή όπως ας πούμε τα στοιχήματα σε ε, κατηγορίες ε, νέων και το στήσιμο στοιχημάτων τέτοιων ομάδων είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ ότι όντως πρέπει αποτελεσματικά να έχουμε μέτρα αντιμετώπισης αυτού του θέματος και πρέπει να έχουμε και πειθαρχία σε επίπεδο ε, αθλητισμού. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συναδελφοί, αλλά νομίζω ότι αυτά ακριβώ αποδεικνύουν ότι όλοι στην ίδια βάρκα βρισκόμαστε και βεβαίως ε, ε, θα συνεργαστώ με μεγάλη χαρά με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σινάλοβα. Να θέσω δύο ερωτήσεις και εγώ. Δύο θέματα που δεν τα κατάλαβα. Μιλήσατε για τα καταχώρηση. Καταχώρηση των ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών ή και των παικτών. Τι εννοείς, Ήβο, όλοι όσοι μπαίνουν σε ένα τέτοιο site καταχωρούνται ή είναι για καταχω... η καταχώρηση αφορά τους, ε, τα site. Την ίδια ερώτηση θέτω προς την Επιτροπή. Εσείς τι λέτε. Ακούσαμε από όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι κρίσιμος. Κομισιόν θα σας δώσω σύντομα το λόγο. Πείτε μου λοιπόν όταν μιλήσετε εσείς τι άποψη έχετε για την προσέγγιση αυτή ότι πρέπει να παίξετε ένα κρίσιμο ρόλο. Πώς το ερμηνεύετε. Ήβο και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πραγματικά μπήκατε στο πιο δύσκολο και πιο κρίσιμο σημείο. Το, έ, το έθεσαν και πολλοί συνάδελφοι. Ο Χάνο, ο οποίος έφυγε. Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν το εθεσαν και πολλοι συναδελφοι ο Χάνου, ο οποιος εφυγε πολλες ιδιωτικες επιχειρησεις που παρεχουν ε, τετοιες ε, δεν είναι καταχωρημένες στην Ένωση. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η καταχώρηση των χρηστών, που είναι βέβαια ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Μιλάμε για έλεγχο στο ίντερνετ και δεν θα υπάρχει πολύ εκτεταμένη υποστήριξη αυτό. Ας προχωρήσουμε προς την άλλη προσέγγιση, την καταχώρηση, τη χορήγηση αδειών, δηλαδή την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή να είσαι υποχρεωμένο να καταχωρηθεί στην Ένωση, είτε είσαι Κινέζο, είτε είσαι οτιδήποτε. Θα πάρει μία άδεια, την άδεια τη δίνει η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή και βέβαια χρειαζόμαστε και ένα εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, γιατί αλλιώ το θέμα είναι άχρηστο. Γιατί εξορισμού πρόκειται για διασυνοριακέ δραστηριότητε. Η προτεραιότητά μα λοιπόν θα πρέπει να είναι να δώσουμε έμφαση στην καταχώρηση και στην αδειοδότηση αυτών των παρόχων υπηρεσιών. Επιτρέψτε μου επίσης, Πρόεδρε, να σχολιάσω κάποιες άλλες προτάσεις που ακούστηκαν από τους συναδέλφους για τα μέτρα, τα κυρωτικά μέτρα, την ε, ποινικοποίηση. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μέτρων στην ανακοίνωσή της, ε, κυρώσεων μπλοκάρισμα των πληρωμών. Εδώ δεν μιλάμε πια για πρόληψη, αλλά για αντιμετώπιση, μπλοκάρισμα των πληρωμών, παρεμπόδιση της πρόσβασης σε παράνομες ή μη καταχωρημένες ιστοσελίδες. Υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα ή τα εφαρμόζουν κάποια κράτη ήδη. Μπορούμε να το κάνουμε σε όλη την Ένωση. Δεν ξέρω. Ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει βέβαια μέσω οδηγίας. Η Κομισιόν προτείνει σύσταση. Εξαιρετικό το κείμενο, αλλά με σύσταση δεν προχωράμε. Μετά, απάτες ε, στα, στοιχήματα, ε, στα αθλητικά στοιχήματα. Εμείς προτείνουμε ενιαίο ενιαίο πλαίσιο κυρώσεων για τις απάτες στα, αθλητής, ε, στα στοιχήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή κάθε κράτος μέλος έχει δική του προσέγγιση. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να υπάρχει μια ομοιόμορφη προσέγγιση της ε, αδικηματικής πράξης. Μιλήσατε για το πολωνικό μοντέλο, τα εισοδήματα δηλαδή από τα τυχερά παιχνίδια να πηγαίνουν στις βασικές, στις τοπικές αθλητικές δομές. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη, αλλά προφανώς μπορούμε να το λάβουμε υπόψη ως μια καλή πρακτική. Για την κυρία Σιλακόβα. Η υπεύθυνη διαφήμιση είναι βασικό στοιχείο της πρόληψης. Δεν μπορεί να μπει αυτό σε οδηγία, αλλά είναι σαφές ότι εδώ η Επιτροπή πρέπει να παράσχει σαφείς ε, ε, καθοδηγητήριες γραμμές μέσω συστάσεων για τον τρόπο λειτουργίας των διαφημίσεων. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να σχολιάσει. Thank you, Madam Chair. Good morning, everybody. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Για τα δύο ερωτήματα ε, που θέσατε. Νομίζω ότι πρέπει και τα δύο να τα εξετάσουμε, να δούμε την καταχώρηση των ιστοτόπων, όπως επίσης και την καταχώρηση του παίκτη. δεν είμαι σίγουρος ότι όλες ε, οι, τυχερε, οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών που είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες μέρες, ε, μέλη μπορούν να ε, καταχωρούνται σε κάθε κράτος μέλος, αν δεν είναι αδειοδοτημένα. Πρέπει να υπάρχει μια αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα τυχερά παιχνίδια. Πρέπει να έχεις και μια αδειοδότηση να προσφέρεις τυχερά παιχνίδια σε μια χώρα. Ε, βέβαια, η καταχώρηση είναι ένας τρόπος ε, προστασίας των καταναλωτών, αλλά επίσης εξασφάλισης του γεγονότος ότι η προσφορά της υπηρεσίας αυτής ε, δεν περιέχει απάτες, ότι δεν θα γίνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όταν, όταν προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες. Ρωτάτε πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Από το 2005 όταν ο Επίτροπος Μπαρνί για πρώτη φορά μίλησε για τα τυχερά παιχνίδια στο Κοινοβούλιο δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε έναν ζωτικό ρόλο, να ηγηθούμε τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύουμε ότι το σχέδιο δράσης παρουσιάσαμε πέρσι τον Οκτώβριο αποτελούσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς μια νέα πολιτική για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Μία φορά να, ακόμη να επαναλάβω ότι είναι ένα πρώτο βήμα και πρέπει να δούμε πόσο επιτυχέ θα είναι αυτό το πρώτο βήμα. Κάποιοι ευρωβουλευτέ είπαν ότι η Επιτροπή μόνο συστάσει προτείνει. Κοιτάξτε, η ήπια νομοθεσία είναι. Δεν είναι μια ισχυρή απάντηση που, ε, που περιμέναμε σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάβαμε υπόψη όλα τα σχόλια. Ε, και για τη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο λάβαμε πάρα πολλά σχόλια. Διαβάσαμε την έκθεση ε, του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι τα πρώτα πράγματα που προτείναμε στο πρώτο σχέδιο δράσης μας είναι ένας καλός τρόπος να κινηθούμε. Γιατί σε εύλογο χρονικό διάστημα θα φανεί αν αυτό το πρώτο βήμα είναι επαρκές για να έχουμε μια, κάποια πλαισίωση των τυχερών παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν αρκεί αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο, να σκεφτούμε περισσότερα και διαφορετικά βήματα. Νομίζω όμως ότι είναι μια καλή αφετηρία για την πολιτική μας αυτή και επίσης ε, είμαι πεπισμένος, ακούγοντας τα μέλη της Επιτροπής σας, ότι μπορούμε να δουλέψουμε επί του πρώτου αυτού βήματος και σε δύο-τρία χρόνια, αν στεφθεί με επιτυχία, βλέπουμε αν χρειάζεται να ε, πάρουμε και περαιτέρω μέτρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ήβο, μήπως θέλεις να πάρεις και πάλι το λόγο. Ναι, απλώς να επιβεβαιώσω ότι αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και σημαντικό δεν είναι το τελικό βήμα και η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι στα ερχόμενα έτη μπορεί να χρειαστούν κι άλλα βήματα και από ό,τι κατάλαβα δεν ε, αποκλείεται το γεγονός Εντάξει, ε, λέτε ότι είναι μια ήπια προσέγγιση, ήπια νομοθεσία. Ναι, αλλά συμπεριλαμβάνει πολύ ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Ας μην ε, έχουμε αυταπάτες. Ε, μπορεί όμως μια ισχυρότερη νομική πρωτοβουλία να είναι απαραίτητη και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχετε την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Να σα υπενθυμίσω ότι η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως θα γίνει το Μάρτιο από τον Ιβο Μπέλεφ και θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μα. Τότε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξή μας ε, για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επιμουσικών οργάνων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή Νομικών είναι η αρμόδια καθήλυν επιτροπή. Εγώ είμαι η συγγήτρια της δικής μας επιτροπής. Θα ήθελα να σας κάνω μία επισκόπηση για το τι βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το σύστημα των ε, συλλογικών, ε, της ε, διαχείρισης, της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων και θα σας πω και ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται συλλογικά τα διαχειρίσματα, των, τα, τα δικαιώματα των δημιουργών οι δημιουργοί μεταφέρουν την διαχείριση αυτή σε, μια, σε έναν ειδικό φορέα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα το μουσικό. Ε, οι εταιρείε συλλογική διαχείρισης υπάρχουν πολλά χρόνια, εδώ και 100 χρόνια περίπου στις περισσότερες κράτη-μέλη, αλλά επειδή υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, ζήτηση για ε, χρήση στο διαδίκτυο των έργων τους ε, έχει, έχει φανεί η ανάγκη ρύθμισης των δικαιωμάτων βάσει των εθνικών φορέων. Η συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων είναι ένας περίπλοκος τομέας γιατί επηρεάζει τη διαχείριση των δικαιωμάτων για επιγραμμική χρήση, αλλά και για χρήση εκτός διαδικτύου, offline. Αφορά τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά και των παραγωγών, των μεταδοτών. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς. Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενή δικαιώματα, αλλά αυτή η οδηγία θα δημιουργήσει ένα ε, περιεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, διακρατικό. Δηλαδή θα ορίσει την νομοθεσία για διακρατική χορήγηση αδειών ε, ε για επιγραμμική χρήση μουσικών έργων. Οπότε όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές συζητήσει ε, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαχείριση των ε, εταιριών αυτών διαχείρισης δικαιωμάτων, ειδικότερα λόγω των προβλημάτων της ψηφιακής συμπεριφοράς πολλών καταναλωτών. Έχουμε μερικά πολύ κακά παραδείγματα. Να πάρουμε το παράδειγμα, για παράδειγμα, μιας εταιρείας ε, στην Ισπανία πρόσφατα υπήρχε απάτη και διαφθορά και ήταν σαφές ότι δεν μπορούν να ε, συνεχίζουν αυτήν την ε, συμπεριφορά τους. Πρέπει να αλλάξουν τη συμπεριφορά, τη διαχείρισή τους. Δεν είναι βέβαια όλες οι εταιρείες αυτές, ε, όλες οι εταιρείες αυτές τόσο κακές στη διαχείρισή τους, αλλά υπάρχει μία συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα σε όλες τις κοινωνίες. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και όπως ήδη είπα είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης του θέματος αυτού. Η προτινόμενη οδηγία έχει δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι η καλύτερη διαχείριση διαφάνεια, δημοκρατική συμπεριφορά στο πλαίσιο των εταιριών ε, για να είναι πιο δημοκρατικές και επίσης οι πληρωμές προς τους δημιουργούς, ε, οι σωστές πληρωμές και έγκαιρες πληρωμές. Όλα αυτά τα οποία δηλαδή θεωρούμε καλή διαχείριση και καλή απόδοση. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα της ε, οδηγίας. Και το δεύτερο τμήμα, ο δεύτερος στόχος αφορά τη διευκόλυνση της ε, διαδικτυακής αδειοδότησης των μουσικών, αγορών, των μουσικών έργων στην ψηφιακή αγορά, δηλαδή αφορά το πώς μπορούμε να έχουμε διακρατική αδειοδότηση για τα μουσικά έργα στο ψηφιακό ευρωπαϊκό ε, περιβάλλον είναι κάτι που το χρειαζόμαστε επιγόντω, ε, γιατί είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Δεν είναι δυνατόν να το ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα εθνικά, όταν το διαδίκτυο υπερβαίνει τα σύνορα ε, των κρατών μελών. Ήδη συζητήσαμε με εμπλεκόμενους φορείς, ε, με εταιρείε συλλογική διαχείρισης ε, και συμφωνούν όλοι με την καλύτερη διαχείριση, τη διαφάνεια, την δημοκρατική λογοδοσία, όπως επίσης και τη διευκόλυνση αυτή της ε, διαδικτυακής χορήγησης αδειών για τα μουσικά έργα. Όταν όμως φτάνουμε σε μερικά περίπλοκα και δύσκολα ζητήματα, θα επικεντρωθώ κυρίως σε αυτά ε, μέσω των τροπολογιών μου. Εκεί τίθεται το ζήτημα, γιατί αν θέλει κανείς μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία, πιο δημοκρατική συμπεριφορά, χρειάζεται βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βάσεις δεδομένων για να μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Και το ερώτημα, είναι, το ζήτημα είναι το εξή ότι έχουμε επίσημες εταιρείες συλλογική διαχείρισης ε, που, ε, και κάποιες χώρες που επένδυσαν πολύ σε αυτό το ψηφιακό εξοπλισμό, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού. Και το κατά πόσο οι εταιρείε αυτές μπόρεσαν ή θα μπορέσουν στο μέλλον να επενδύσουν σε αυτό το ψηφιακό τους εξοπλισμό, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατόν ε, να έχουν πολύ καλή διαχείριση. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει στο επόμενο ερώτημα, ποια είναι η σχέση μεταξύ πολύ αποτελεσματικών ε, εταιριών και λιγότερο αποτελεσματικών εταιριών διαχείρισης. Ε, μπορεί να είναι μεγάλες εταιρείε που είναι πιο αποτελεσματικές, μικρότερες που είναι λιγότερο αποτελεσματικές, μεγάλες, χώρες, ε, μεγάλες εταιρείε στις δυτικές χώρες και μικρότερες στις ανατολικές χώρες με περισσότερα προβλήματα. Οπότε τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Πώς θα συνεργαστούν και πώς θα τα καταφέρουν. Και να πάω τώρα στο επόμενο σημείο, γιατί επιχειρηματολογεί η Επιτροπή ότι κάποιες από τις επίσημες εταιρείες ε, θεωρούν ότι ολόκληρη η οδηγία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία, γιατί Υπάρχουν ορισμένα ρεπερτόρια που ε, στρέφονται προς συγκεκριμένους ε, ακροατές ε, και αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί καλύτερα. Υπάρχουν άλλες εταιρείες διαχείρισης που λένε ότι όχι, δεν νομίζουμε ότι θα γίνει αυτό. Ίσως το θέμα φορά περισσότερο το ευρύτερο ρεπερτόριο και όχι το πιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Αν υπάρχει πρόβλημα με το μικρότερο ρεπερτόριο και απειλείται κάποιο είδους ρεπερτόριο, ε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης και προσβασιμότητας ε, του πιο μικρού, πιο συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Κάτι ακόμη στο οποίο θα επικεντρωθώ είναι ο θεμητός ανταγωνισμός η ιδέα της Επιτροπής είναι καλός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών διαχείρισης των ε, δικαιωμάτων και των τριών πλατφορμών. Δεν θέλουμε δηλαδή μονοπόλια εταιριών συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να γίνει η διαδικτυακή χορήγηση άδεια αν υπάρχει αυτή η ψηφιακή βάση για την οποία μίλησα. Όμω πρέπει να υπάρχει και μια σαφή νομοθεσία για τι εταιρείε συλλογική διαχείριση ε, και ε, για, την, για τις πλατφόρμες επιλογής 3 να αναρωτηθούμε αν αφορά όντως τον ανταγωνισμό ή αν στο μέλλον πρόκειται να υπάρξει ε, άνηση ε, εξέλιξη των ε, εταιριών συλλογική διαχείρισης, δηλαδή μεγαλύτερη ρύθμιση για μερικές εταιρείες και μικρότερη ρύθμιση για κάποιες άλλες. Ο θεμητό ανταγωνισμό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα και θέλω να είναι η ισότιμη κατάσταση για όλους του εμπλεκόμενου φορεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξασφαλίσουμε και σε αυτό θα επικεντρωθώ κυρίως από την άλλη αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βέβαια πολύ λεπτομερές και είναι πολύ καλή δουλειά ε, και μια πολύ καλή πρόταση αυτή που μας υπέβαλαν και βεβαίως θέλουν να έχουν τη δυνατότητα αν ένας δημιουργός δεν μπορεί να βρει μια εταιρεία που να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του ε, ή να δώσει άδεια μπορούν, μπορεί να πάει σε μία άλλη ε, εταιρεία ή σε έναν άλλο φορέα ή να μπορεί να το κάνει μόνος του. Να υπάρχουν δηλαδή και πιο ε, μεμονωμένες επιλογές για το δημιουργό, κάτι το οποίο για μένα είναι θετικό μάλλον. Τέλο πάντων, είναι πολύ καλέ ιδέε και πολύ καλή δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω υπάρχουν τρία μεγάλα ζητήματα. Για τον εξοπλισμό, στον εξοπλισμό αναφέρομαι και τη δυνατότητα ανάπτυξή του το θέμα της ε, πολιτιστικής ε, ε, ποικιλομορφία και το θέμα της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και την καλή ρύθμιση των εταιριών συλλογικής διαχείρισης και τους κανόνες δίκαιου ανταγωνισμού. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου και θα ήθελα συνεπώς να σας καλέσω να πείτε τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Χέλγα. Πολλά από αυτά που είπες ε, μπορώ να τα υποστηρίξω 100%. Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή θα βρούμε μια κοινή γραμμή. Ήθελα να τονίσω ότι η βασική προσέγγιση της Κομισιόν για, τον, ε, για τις συνθήκες του δικαίου ανταγωνισμού και τις ίδιες συνθήκες για όλες τις εταιρείες αυτές ε, για όλη την Ευρώπη και που θέλει δηλαδή και νομικός να το αριθμίσει είναι νομίζω μια λογική προσέγγιση. Το βλέπουμε ότι σε πολλές εταιρείε αξιολόγησης υπάρχει μεγάλος βαθμός αδιαφάνειας και οι καλλιτέχνε συνεργάζονται με τέτοιε εταιρείε και πολλέ φορέ δεν είναι ικανοποιημένοι γιατί δεν μπορούν πάντα να ξέρουν αν όντω ο τρόπο που υπολογίζουν οι εταιρείε αυτέ όσα υπολογίζουν είναι ο σωστό ή ο συμφέρον για του καλλιτέχνε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει όντω ένα θεμητό ανταγωνισμό και αυτό είναι λογική και σκόπιμη προσέγγιση. Νομίζω ότι πολλά από τα σημεία που υπάρχουν στην πρόταση τη Κομισιόν αξίζει να, υποστηριχθούν, είναι λογικά. Σημειώνω, ή μάλλον έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποια σημεία όπου υπάρχει μια ανισορροπία στην πρόταση της Κομισιόν. Από τη μία δηλαδή είναι πολύ λεπτομερής η αναφορά για το τι γίνεται με τις εταιρείε συλλογική διαχείρισης, ε, ποια είναι τα δικαιώματα των μελών τους κτλ. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερέστατα και μπορούμε να το συζητήσουμε αν όντως χρειάζεται και αυτός ο βαθμός λεπτομέρειας. Από την άλλη, κεντρικά θέματα, βασικά θέματα ε, δεν τη τις ίδιες λεπτομέρειες. Ας πούμε, αν υπάρχει μια υποχρέωση ε, συγκεκριμένων τελών, ε, τι γίνεται με το πώς αναλαμβάνει μια τέτοια εταιρεία, τη διαχείριση. Όλα αυτά δεν είναι απολύτως σαφή. Ίσως λοιπόν για κάποια σημεία να πρέπει να, να υπάρξει έτσι μια μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης έχω την εντύπωση ότι ε, η, λέει η πρώτης Κομισιόν ότι αυτές οι εταιρείε συλλογική διαχείρισης ε, οργανώνονται στα κράτη-μέλη ε, με τον ίδιο τρόπο περίπου ε, ότι δηλαδή οργανώνονται από, σαν εταιρείε μελών. Ε, αν αυτές οι εταιρείε αν αυτές τις διαχείρισης θέλουμε να τι ε, ε, ρυθμίσουμε, το θέμα είναι τι θα γίνει με τις υπηρεσίες αδειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξάνονται συνεχώς και τι κάνουμε και με τους μεγάλους παίκτες επίσης, στον τομέα της μουσικής για παράδειγμα που δεν υπόκεινται σε αυτέ τι εταιρείε συλλογική διαχείριση. Θα του διαχει... θα τους θεωρήσουμε το ίδιο με τι εταιρείε συλλογική διαχείριση. Δηλαδή, όντω δημιουργούμε έναν θεμητό ανταγωνισμό ή μήπως δημιουργούμε ένα σύστημα όπου αυτές οι εταιρείες ε, διαχείρισης ε, ρυθμίζονται πάρα πολύ αυστηρά και από την άλλη κάποιες υπηρεσίες ή εταιρείε ε, αδειοδότησης ή οι μεγάλοι, παίκτες στην αγορά του, της μουσικής την χάνουν πιο ευέλικτης έτσι, αντιμετώπισης. Πρέπει να δούμε και το θέμα της προσβασιμότητας για τα διάφορα είδη ας πούμε μουσικής. Ε, νομίζω ότι ε, αν ε, θα ήταν προβληματικό να δημιουργηθεί, θα ήταν μάλλον δύσκολο ή θα ήταν και ίσως αδύνατο να δημιουργηθεί αυτός ο θεμητός ανταγωνισμός με αυτές τις συνθήκες. Οπότε ερώτημα προς την Κομισιόν. Εσείς με αυτές τις εταιρείες αδειοδότησης που υπάρχουν παντού στην Ευρώπη, πώς ακριβώς θέλετε να προχωρήσετε θα πρέπει και αυτές να υπόκεινται στις ρυθμίσεις, τους κανόνες για τις εταιρείε συλλογική ε, συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, ένα ακόμα ερώτημα για, τον δεύτερο, για το δεύτερο κομμάτι της οδηγίας, για την ε, online μουσική και την παροχή online μουσικής. Ε, τι γίνεται με τις άδειες. Ε, τίθεται και εκεί το ερώτημα. για ε, αδειοδότηση διασυνοριακή όλοι υποχρεούνται να υπόκεινται σε αυτές τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι ουσιαστικά και το ερώτημα που έθεσα και πιο πριν. Ε, γιατί πάντα διαπιστώνω ότι για τους μεγάλους παίκτες ε, οι κλασικές ας πούμε εταιρείες ε, συλλογική διαχείρισης είναι πολύ περίπλοκες, δεν είναι πολύ ελκυστικές, θέτουν σε εμπορία τη μουσική περισσότερο από μόνοι τους και όταν κάποιο θέλει ας πούμε, να ακούσει μουσική στο ραδιόφωνο ή στο ίντερνετ ή στο τηλέφωνό του ή οπουδήποτε αλλού, ε, δεν υπάρχουν πάντα οι δυνατότητε ε, τόσο. σω να πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία θηρίδα ε, για, για να μπορεί κανεί να ζητήσει, ας πούμε, μια άδεια για να παρέχει μουσική. Τώρα το αν θα έχουμε μεγάλες ας πούμε συμπράξεις τέτοιων εταιριών ε, στην Ευρώπη ή θα έχουμε κάτι άλλο είναι, ε, δεν είναι ε, σημαντικό. Σημαντικό είναι να έχουμε τη δυνατότητα για τέτοιες άδειες για μουσικές εταιρείε να μπορεί κανείς να, ζητήσει, να τις ζητήσει και διασυνοριακά, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα και τα βασικά προβλήματα μια, ε, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με μια τέτοια οδηγία είναι να υπάρχει πιο εύκολα, ε, πιο, να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες και πιο εύκολες ε, ε, συνθήκες ώστε να μπορεί κανείς να ζητήσει, να λάβει, να χρησιμοποιήσει μουσικά κομμάτια. Για τον χρήστη λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες, ε, περισσότερες μάλλον ευκαιρίες ανεξάρτητα από το πού προέρχεται αυτή η, ε, η μουσική. Ε, και βεβαίως όλες αυτές οι περαιτέρω δυνατότητες θα πρέπει να είναι προφανώς νόμιμες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της πειρατείας. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά ερωτήματα που ακόμα έχουν μείνει εκκρεμή. Η βασική αρχή, η βασική προσέγγιση είναι καλή και φαντάζομαι ότι εδώ αυτή την καλή προσέγγιση θα την συνεχίσουμε, θα την βελτιώσουμε στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε στο τέλο να καταλήξουμε να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε έναν θεμητό ανταγωνισμό, να έχουμε ίδιε συνθήκε για όλου και πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρα. Ο κύριο Σεγκάλσκι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πω ποια είναι η άποψη της ομάδας μου, του ECR. Ε, η συνάδελφοι που ήταν υπεύθυνη ήταν στην ΙΜΚΟ και θα διαβάσω τι μου ετοίμασε. Υποστηρίζουμε τους δύο στόχους που υπέβαλε η Επιτροπή για τη βελτίωση της διακυβέρνησης ε, των ε, εταιριών διαχείρισης και ενθαρρύνουμε για να διευκολύνουμε τη χορηγήση πολλαπλή εδαφική ισχύω αδειών για online χρήστε. Υποστηρίζουμε τι μεθόδου για την απλοποίηση και βελτίωση της αδειοδότησης των online έργων και καλωσορίζουμε πολλά από όσα περιλαμβάνει το σχέδιο οδηγίας. Θα δουλέψουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τα κείμενα εξασφαλίζει την, ε, τις του streamline ε, και για την υπέρβαση εθνικών εμποδιών που μπορεί να υπάρχουν για την απαγόρευση τέτοιων ε, εμπορικών φορολογικών ρυθμίσεων, ώστε αυτέ να είναι και ελκυστικέ και κοστοποτελεσματικέ για όσους ζητούν να πάρουν άδεια για έργα για online χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν τομεί ανησυχία από πλευρά μας. Πολλά θέματα μπορούν να βελτιωθούν για να διευκολύνουν τις τάξεις, για να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση με τις καλές πρακτικές ιδίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνάδελφος προτείνει μια σειρά τομέων να εξετάσουμε. Πρώτον, ο ορισμός της εταιρεία διαχείρισης συλλογικών ε, δικαιωμάτων στο άρθρο 3 στηρίζεται σε οργανώσεις που στηρίζονται σε μέλη. Δεύτερον, η πρόταση, τα κονδύλια που συλλέγονται αλλά δεν μπορούν να συντεριαστούν να διατηρούνται από τις εταιρείε ε, μετά από μια περίοδο 5 ετών. Άρθρο 12. Μας ανησυχεί. Αυτό είναι το ανάποδο από αυτό που έχει σαν βασική θέση το Ηνωμένο Βασίλειο και αντικατοπτρίζεται στην εθνική νομοθεσία. Το Αυτή είναι η θέση της κυρίας Μακλάρκ. Επίσης, και μου ζήτησε να την ε, ε, επαναλάβω, να την παρουσιάσω εδώ. Προφανώ θα δουλέψει για το θέμα αυτό από εδώ και στο εξή, οπότε νομίζω ότι καλό είναι να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκάλσκι, παρουσιάζοντας τις απόψεις της κυρίας Μακλάκλιν. Ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ. Ε, Νομίζω ότι η εναρμόνιση του συστήματος αυτού είναι εξαιρετικά καλή. Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε συγκεκριμένες, τις συγκεκριμένες δομές τα, σε διάφορα κράτη-μέλη, γιατί δεν είναι αναγκαστικά ε, μια νομική διαδικασία γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να υπάρχει λοιπόν εσωτερική διαφάνεια, ιδίως σε ό,τι αφορά το, την εσωτερική λειτουργία αυτών των δομών. πρέπει να λάβουμε υπόψη ωστόσο κάποια ζητήματα. Υπάρχει στην Πολωνία μία ένωση πνευματικής ιδιοξίας που έχει ηλικία άνω των 100 ετών, έχει... δεν είναι συσσωματίου, μία μη κυβερνητική οργάνωση είναι στην πραγματικότητα, έχει διαχειριστεί χιλιάδες έργα χιλιάδων συγγραφέων και λειτουργεί μια χαρά το σύστημα. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Βέβαια, η διαφάνεια είναι σημαντική, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συγκεκριμένα συστήματα των κρατών μελών. Συχνά τα συστήματα αυτά λειτουργούν μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων, οργανώσεων. Τα χρήματα λοιπόν που κερδίζουν επενδύονται σε συστήματα καλύτερης διαχείρισης online ε, των έργων αυτών. Συχνά μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες μουσικής, ε, τέχνης ή γλώσσας και είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες που έχουν η ειδική αυτή δημιουργεί. Αν επιβάλλουμε το ίδιο σύστημα σε όλους, θα δυσκολευτεί η λειτουργία των μικρών και μεσαίων φορέων. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι δομές. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Μπόρις. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Η κυρία Πράτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τη λεπτομεριακή παρουσίαση και σχολιασμό των μελών. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Θα σταθώ σε δύο-τρία θέματα και μετά θα σχολιάσω κάποια από τα σχόλια των βουλευτών. Να τονίσω την ανάγκη της πρότασης και τους λόγους για τους οποίους υποβάλαμε την πρόταση αυτή. Πρώτον, διότι πιστεύουμε ότι οι οργανώσεις συλλογική διαχείρισης των δικαιωματοφτών έχουν βασικό ρόλο στο σύστημα της διαχείρισης του copyright δεν υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια όπως αναφέρθηκε πάντα, αλλά θέλουμε να το κάνουν ε, με σωστό τρόπο στον 21ο αιώνα. Όταν άλλαξε ο τρόπος εξμετάλλευσης, όταν άλλαξαν οι εμβέλειες των παρόχων, όταν η ανάγκη της διαφάνειας είναι μεγαλύτερη. Και σωστά το το, το, το ζητούν. Ωστόσο η Επιτροπή δεν θέλει να δυσκολέψει τη ζωή των δομών αυτών, αλλά για να κάνει ουσιαστικό το αποτέλεσμα της δουλειά τους. Σκεφτείτε ότι μία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης στην Ευρώπη δεν εκπροσωπεί μόνο τα μέλη της, αλλά όλους τους δημιουργούς στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια και δεν πρέπει αυτή τη διαφάνεια να την βλέπουμε μόνο από την οπτική γωνία των μελών αλλά και από την οπτική γωνία των άλλων μελών στα άλλα κράτη. Και, και είναι αναγκαίο και για τους ε, χρήστες. Κάποια από τα δικαιώματα και κάποιοι από τους δικαιούχους ε, συχνά δεν μπορούν να, τύχουν, να λάβουν τις άδειε που χρειάζονται. Και αυτό εν τέλει επιβαρύνει τον καταναλωτή, τον Ευρωπαίο πολίτη. Κύριε Τρίπελ, τρία θέματα θέσατε ως σημαντικά για τα οποία ζητήσατε την άποψη της Επιτροπής. Πρώτον, τεχνικές δυνατότητες, ιδιαίτερα για τις online άδειε και αν αυτό μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες ή τις αποτελεσματικές εις βάρος των μη αποτελεσματικών όπως το είπατε. Πρώτον, η απέτηση να υπάρξουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, που είναι κάτι που ήδη συμπεριλάβαμε για την, την χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύω, είναι ουσιώδου σημασίας και είναι και δυνατό. Δεν μπορεί πλέον να έχουμε εταιρείε που δεν μπορούν να πούν στους χρήστες τι αδειοδοτούν και να μην διανέμουν στους δικαιούχους τα δικά τους λεφτά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτές οι τεχνικές ε, απαιτήσει που δεν υπήρχαν στο παρελθόν για τους χρήστες απαιτούνται τώρα, διότι απαιτούνται για την μορφή αυτή της ψηφιακής εκμετάλλευσης και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε μερικές μικρές εισαγωγικά επιχειρήσεις που έχουν εξαιρετικά καλές επιδόσεις και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τόσο καλά. Δεν είναι λοιπόν μια μάχη μικρών μεγάλων, αλλά μια προσπάθεια να επιτρέψουμε σε όλους να λειτουργήσουμε κάποια minimum απαιτούμενα standard. Και δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι επενδύσεις ή να ακολουθηθούν από όλες τις εταιρείες συγκεκριμένες τεχνολογίες. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να έχει το γραφείο διεκπαιρέωσης εκτός ε, της εταιρείας για να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή την τεχνική δυνατότητα που απαιτείται. Αυτό συμβαίνει ήδη, απλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα το κάνουν όλοι. Δεν επιβάλλουμε ωστόσο τούτο ως τον μόνο τρόπο λειτουργίας των ε, εταιριών συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ δυνατότητες και βεβαίως περιλαμβάνουμε την υποχρέωση να γίνει δεκτό το κόλλημα, η συγκόλληση, η συνένωση, το tagging on των διαφόρων μικρών εταιριών. Αυτό το βλέπουμε ήδη στο άρθρο 29 και 30 της οδηγίας. Το δεύτερο θέμα σας, κύριε Τουίπελ, η ανάγκη να υπάρχει ένα ευρετήριο εχμής, το νήσο ρεπερτουάρ. Οι εταιρείε αυτές συλλογικής διαχείρισης είναι ε, χρήσιμες για να προωθήσουν στην αγορά και ένα ρεπερτόριο που δεν θα είναι τόσο εμπορικό αλλά θα εκπροσωπεί και άλλες τάσεις. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για σας, αλλά και για τον πολίτη και για τους ίδιους τους παρόχους. Αν δείτε τις λίστες των ε, μουσικών ε, έργων online, θα δείτε ότι εκεί η πολιτιστική, η μουσική διαφοροποίηση είναι καλύτερα παρουσιασμένη εκεί από ό,τι στα μαγαζιά. Έχουμε έναν κατάλογο με 30 εκατομμύρια μουσικά έργα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μαγαζιά δεν τα δίνουν όλα αυτά. Και γιατί, διότι υπάρχουν πολίτες που θέλουν το τοπικό ρεπερτόριό τους. Σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία θα δείτε ότι 50% περίπου της μουσικής που παίζεται είναι τοπικής παραγωγής ή ντόπιων καλλιτεχνών. Και είναι λάθος να νομίζουμε ότι μόνο τα αγγλοαμερικάνικα είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους παρόχους, μικρούς ή μεγάλους. Και ακριβώς λόγω του ότι θέλουν να έχουν πρόσβαση στο τοπικό ρεπερτόριο, χρειάζονται βελτίωση στην διαχείριση αυτών των συλλογικών, τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Και κάτι ακόμα. Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων και νέων υφιστάμενων δομών και νέων πλατφορμών διαχείρισης αυτές οι πλατφόρμες όλες συνεργάζονται με τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Δημιουργήθηκαν μετά από πρωτοβουλία των ε, μουσικών παραγωγών που δεν είναι όμως το χώρο της ε, συλλογής των, πνευματικών δικαιωμάτων. που παρέχουν τις υπηρεσίε αυτές και έχουν δημιουργήσει τις πλατφόρμες. Εμείς αυτή την πραγματικότητα τη λαμβάνουμε υπόψη και θέλουμε να παρέχουμε τους ίδιους κανόνες Το βλέπετε και στο άρθρο 31 της οδηγίας αυτό. Ακούσαμε σχόλια για το, το βαθμό λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνει η οδηγία, το συζητούμε ακόμα. Κάποιοι λένε ότι παρά είναι λεπτομεριακή, λεπτομερής η οδηγία, άλλοι λένε ότι δεν έχει επαρκείς λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια σωστή ισορροπία, λαμβάνοντα υπόψη ότι και αυτοί, αυτές οι οργανώσεις συλλογική διαχείρισης έχουν διαφορετικό νομικό καθεστώς από χώρα σε χώρα. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, ο χώρος ε, των εταιριών συλλογική διαχείρισης είναι τεράστιος και διαφοροποιημένος. Έχει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, φερειπίν τις εταιρείε των συγγραφέων που έχουν συχνά τη διαχείριση αποκλειστικών δικαιωμάτων. Έχουμε οργανώσεις που είναι μόνο πλατφόρμες, αμπομπρέλες ε, συλλογικέ επιχειρήσεις, ε, εταιριών με μέλη. Π.χ η ε, σωστή αποζημίωση ιδιωτικών αντιγράφων. Έχεις, έχει άλλες περιπτώσεις, υβριδικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι όλοι καλλιτέχνες, συγγραφείς, ε, ε, ερμηνευτές. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση χωρίς να την αλλάξουμε ιδιαίτερα ή να, την, να παρεύουμε σε αυτές. Κάποιοι έφυσαν το ερώτημα γιατί δεν επεκτείνουμε τους κανόνες της οδηγίας πέραν της οδηγίας. Προσέξτε, εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των εταιριών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, όχι να επιβάλλουμε, γιατί αυτό θα έχει και νομικές επιπτώσεις για την λειτουργία των ατομικών ε, δικαιούχων ένα, μια τηλεοπτική, ένας τηλεοπτικός σταθμός, ένας σταθμός εκπομπής δεν κάνει συλλογική διαχείριση αλλά πληρώνει. Δεν έχει στόχο η οδηγία να λέει στις, ε, σταθμού ε, στους σταθμούς πώς θα αντιμετωπίσουν την καταβολή ή την πληρωμή των δικαιωμάτων. Ο λόγος που παρενέβημεν, ιδίως στον τομέα των αδειών πολλαπλής εδαφικής χρήσεως είναι διότι οι χρήστε αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια προβλήματα. Όταν θέλουν να πάρουν τα δικαιώματα όχι από ατομικούς δικαιούχους αλλά από εταιρείε συλλογική διαχείρισης. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και η οδηγία, αυτό είναι πολύ σαφές, δεν θέλει να πάει παραπέρα από τη διαχείριση, συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Άλλα σχόλια που έγιναν από την ECR, αν κατάλαβα το όνομα της κυρίας Κλάρκ σωστά, για το άρθρο, το 12 και 13. Νομίζω ότι δεν το καταλάβατε καλά. Δεν είναι, αυτό, δεν είναι άδεια της συλλογική, της εταιρείας να κρατήσει τα δικαιώματα, τα χρήματα, κονδύλια, αλλά ε, ότι επιβάλλουμε υποχρέωση στην εταιρεία να διανύμει με επιμέλεια και ταχύτητα τα χρήματα. Όταν δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτό, που θα πρέπει να είναι πολύ μικρό ποσοστό στις κανονικές συνθήκες, και θα είναι δικαία. Το, αν το ποσοστό είναι υψηλό θα δείχνει ότι δεν λειτουργεί καλά η εταιρεία αυτή. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να διανεμηθούν τα κονδύλια, πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν κλπ. κλπ για να βρουν τους δικαιούχους, αλλά τότε να αποφασίσουν τι γίνεται με τα κονδύλια. Οι δικαιούχοι είναι, όχι οι εταιρείε συλλογική διαχείρισης. Οι δικαιούχοι λένε τι θα γίνουν τα κονδύλια αυτά μπορεί να πάει σε ένα ταμείο ολοβοήθεια, δεν ξέρω. Αλλά δεν, εμείς απλά προσπαθούμε να μην δώσουμε, να πούμε τι θα γίνει με τα χρήματα, όχι να δώσουμε δικαιολογίες στις επιχειρήσεις για να κρατήσουν τα χρήματα. Αυτά. Είμαστε βέβαια στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Ευχαριστώ την κυρία Πράτ. Νομίζω ότι αποκτήσαμε έτσι μια γενική εικόνα για το ποιοι είναι οι προτινόμενοι στόχοι της οδηγίας και βεβαίως ε, μας αιτιολόγησε και η Κομισιόν την ε, δική της πρόθεση με όλα αυτά που προτείνει, με τις διάφορες παραγράφους. βέβαια οι ανησυχίες που είχαν ε, ανακύψει στην ε, συνεδρία της προηγούμενης εβδομάδας με τους εκπροσώπους του κλάδου δεν έχουν καλυφθεί απολύτως. Το είπε και η Πέτρα ε, και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπες ε, Πέτρα. Ας δούμε λοιπόν τα σημεία που ακούστηκαν και σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως η... όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για να βελτιωθεί η οδηγία, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τίποτα. Όλοι είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι, ξέρουμε ότι υπάρχει ψηφιακή αγορά, θέλουμε να υπάρχουν νόμιμες προσφορές, θέλουμε ο... οι χρήστες να είναι νομικώς εξασφαλισμένοι, αλλά να, και οι δημιουργοί να μπορούν να ε, είναι και αυτοί εξίσου εξασφαλισμένοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή διαχείριση για να δούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την λειτουργία των εταιριών αυτών συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων. Θα κάνουμε λοιπόν ε, τις προτάσεις μας τον Απρίλιο στη συνεδρίασή μας θα έχουμε τις προτάσεις, τον Ιούνιο θα ψηφίσουμε και πόσο ξέρουμε η η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο πριν τις ε, καλοκαιρινές διακοπές έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε και στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας που έχουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις, για τις παρεμβάσεις, για τα σχόλια και βεβαίως τις επόμενες εβδομάδες θα τα ξανασυζητήσουμε όλα. Πάμε τώρα παρακάτω και Συνεχίζω στα αγγλικά. Πάμε στο σημείο 6. Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία σύντομη παρουσίαση από τον κύριο Αλφόνση για τις γενικές γραμμές της εκθέσεως πρωτοβουλίας του, για τις ε, γλώσσες που απειλούνται σε, με εξαφάνιση και για τη γλωσσική πολυμορφία. Η εξαφάνιση των διαφόρων γλωσσών δεν είναι καινούρια. Από αρχαιότητα των χρόνων ε, διάφορες γλώσσες πεθαίνουν. Υπάρχουν ε, όμως πολύ ανισχυτικοί ρυθμοί εξαφάνισης ευρωπαϊκών γλωσσών σήμερα. 7.000 γλώσσες υπάρχουν σήμερα, 3.000 βρίσκονται υπό εξαφάνιση και κάποιες θα εξαφανιστούν Όντω, εάν τα προγράμματα τα ε, προστασίας τους δεν εφαρμοστούν σωστά. Ο κύριο Αλφόνση επικεντρώνει την προσοχή του σε αυτό, προσπαθεί να τονίσει όχι μόνο τον λόγο για τον οποίο όλες αυτές οι γλώσσες ε, ε, απειλούνται στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη, αλλά και τι πρέπει να γίνει για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να διατηρήσουμε και την πολιτιστική και την γλωσσική κληρονομιά τη Ευρώπη. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Αλφόνση. Ευχαριστώ πολύ. Όλες οι γλώσσες της Ευρώπης είναι σημαντικές για τη ταυτότητά της ε, και στην Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες γλώσσες ε, και κάθε μία από αυτές ε, είναι σημαντικό τμήμα της ε, πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης. Υπάρχει και μία επιστημονική προσέγγιση γιατί η UNESCO άρχισε πρώτη να μιλάει για αυτό το θέμα. Μία διάγνωση της υγείας των γλωσσών βάσει κάποιων κριτηρίων της μεταλαμπάδευσης της γλώσσας από τη μία γενιά στην άλλη, τη χρήση από τους διάφορους ομιλητές ομιλητές της γλώσσας, όπως επίσης και διαφόρων τεχνικών κριτηρίων ε, σε σχέση με την εκμάθηση και, τον, ε, και τις μεθόδους, ε, τους τρόπους εκμάθησης. Αυτή η διάγνωση δίνει τη δυνατότητα σήμερα να πούμε με βεβαιότητα ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές δεκάδες γλώσσες οι οποίες απειλούνται είτε περισσότερο είτε λιγότερο με εξαφάνιση. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο παρελθόν ε, εδώ και 30 χρόνια είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με τις ε, γλώσσες τις μειονοτικές. Είναι τμήμα της πολιτιστικής, αυτό, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια αυτή ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας χάρτης μειονοτικών γλωσσών της Ευρώπης. Έχει λοιπόν ένα θετικό ρόλο διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν και πρέπει να αναλάβει εκ νέου αυτό το ρόλο σήμερα, γιατί τα τελευταία χρόνια η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και παρατηρείται όχι μόνο επίσπευση της αλλίωσης της πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης, αλλά και μια χαλάρωση στις δημόσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, γιατί η γλώσσα είναι μια κληρονομιά της κοινότητα που την ομιλεί, αλλά είναι και μια κληρονομιά ευρύτερη για την Ευρώπη. Ε, τα Κορσικά, για παράδειγμα, η γλώσσα της ε, ε, περιοχής από την οποία έρχομαι εγώ, ψικάνικα είναι ε, ένα τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς Ευρώπης. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα καθήκον, μια αποστολή να επαγρυπνά για το θέμα αυτό των γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφία. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ε, όφελος, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ικανότητας της Ευρώπης, ε, ε, της ικανότητας δράσης και προσέλκυσης ε, ε, επισκεπτών, όπως επίσης και παραγωγής πολιτιστικής, ε, γιατί βάσει αυτής πολιτιστικής ε, ποικιλομορφία αυξάνουμε τα θέματα, τη θεματολογία των καλλιτεχνικών μας δημιουργημάτων. Κάτι που στη συνέχεια βέβαια δείχνει την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης. Υπάρχουν βέβαια χώρες οι οποίες έχουν εξαιρετική πολιτική όπως η Φινλανδία ε, η γλώσσα των Σάμι εδώ και ε, πολλά χρόνια ε, είναι αντικείμενο μιας πολιτικής προώθησης. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χώρες οι οποίες δεν δέχονται την πολιτιστική ποικιλομορφία που υπάρχει στην επικράτειά τους, δυστυχώς, και πρέπει κάποια μέρα να τιμήσουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη και κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολιτική για τις απειλούμενες γλώσσες, ε, γιατί η πολιτιστική κληρονομιά ε, απειλείται επίσης μέσω της απειλής ε, κατά των γλωσσών αυτών είναι μια ευθύνη την οποία επιβεβαίωσε εκ νέου η συνθήκη της Λισαβόνας ε, γιατί η γλωσσική ποικιλομορφία είναι σημαντικό τμήμα και βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταρχάς να διαδίδει τις σωστές πρακτικές σαν αυτή της Φινλανδίας οι οποίες πρέπει κατά τη γνώμη μας να ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαγρυπνά προκειμένου οι καλές πρακτικές να ε, διαδίδονται ώστε να μπορέσουμε να διαιωνίσουμε την ευρωπαϊκή μας πολιτιστική κληρονομιά. Τώρα, ως προς, ως προς, το... προς εμάς το Κοινοβούλιο, ε, και πάλι πρέπει να ε, αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση γιατί στα τελευταία δέκα χρόνια όπως είπα η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγη προσοχή έδωσε ε, και λίγο πίεσε την Επιτροπή σε σχέση με το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιβράδυνση τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά και των κρατών μελών που έχουν την πρώτη ευθύνη για το θέμα αυτό και πρέπει να βρούμε τη διατύπωση και τα μέσα να πείσουμε τους υπεύθυνου ε, αποφάσεων ότι πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Δεν ισχύει πάντοτε βέβαια αυτό. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει και ένα θέμα μεγέθους γιατί μια μικρότερη κοινότητα μπορεί να έχει λιγότερη δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα. Τέλος πάντων είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, κάτι το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε στην έκθεση αυτή. Ποιο είναι ο στόχο, θα αρχίσει μια νέα περίοδο πολιετού προγραμματισμού, 2014 με 2020, και πρέπει να ανανεώσουμε την πολιτική μας βούληση και το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των ε, ε, μειονοτικών γλωσσών ε, και να μην παραγνωριστεί αυτό το θέμα όπως έγινε και ήταν ο μεγάλος σαπών η γλωσσική ποικιλομορφία στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι κοινωνίες αυτές οι οποίες έχουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά γιατί οι πληθυσμοί που την κληρονόμησαν από τις προηγούμενες γενναίες ε, έχουν μια συγκεκριμένη πολιτιστική δράση. Πρέπει αυτές λοιπόν οι κοινότητες να ε, ενθαρρυνθούν ε, και αυτό χρειάζεται μια καλή πρακτική. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη-μέλη, πρέπει να ε, επενεθούν αυτές οι γλώσσες να προωθηθούν, ε, ειδικότερα στις χώρες όπου δεν γίνεται αυτό, για να τους δείξουμε τι πολιτικό σφάλμα είναι αυτό για μια μεγάλη ευρωπαϊκή δημοκρατία να μην λαμβάνει επιπλέον υπόψη ε, την μεγάλη γλωσσική ποικιλομορφία που υπάρχει στην έδαφος της. Ευχαριστώ πολύ, Φρανσουά. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Uh, Εντάξει. Να δώσω τότε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το θέλει. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές ε, περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Όχι μόνο αυτές όμως. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, Όλες οι γλώσσες σχεδόν στην Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται σε κίνδυνο με βάση αυτή τη μελέτη της Metanet για την ψηφιακή υποστήριξη των γλωσσών και τα γερμανικά που είναι η περισσότερο μιλούμενη γλώσσα δεν υποστηρίζεται πλέον πλήρως ε, ψηφιακά. Το πρόβλημα υπάρχει λοιπόν. Υπάρχουν προφανώς φαινόμενα που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση της, της οικονομίας, τη διεθνοποίηση κάθε δραστηριότητα στην κοινωνία μας, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις γλώσσες. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο προφανώς και τις μικρότερες και είναι δύσκολο για τις γλώσσες αυτές να ετοιμαστούν έργα που μπορεί να λάβουν χρηματοδότηση από τους, τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να βρουν τρόπους συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ζητήσουν κονδύλια ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα επιβαρύνεται από ένα άλλο φαινόμενο. Τον τον αναλφαβητισμό που αντιμετωπίζουν οι γλώσσες, όλες οι γλώσσες. Ο αριθμός των αναλφαβήτων στην Ευρώπη αυξάνεται, αντί να μειώνεται. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για όλες τις γλώσσες. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες όλες τις γλώσσες που πάνω, βρίσκονται σε κίνδυνο μέσω των προγραμμάτων για εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και με άλλες δράσεις στον τομέα της έρευνας στην ε, Γενική Διεύθυνση πληροφορία, ε, κοινων, ε, της Κοινωνίας υπάρχουν προγράμματα για όλες τις γλώσσες από την ε, ε, τις, τις γλώσσες των μεταναστών, τη γλώσσα των κοφαλάλων, παρότι η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα συγκεκριμένη στον τομέα των περιφερειακών γλωσσών, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Φρανσουά, θες κάτι? Όχι. Βεβαίω να συναντήσω την Επιτροπή και να συζητήσω μαζί τους. Πιστεύω ότι κάθε γλώσσα δεν είναι το θέμα, το θέμα δεν είναι το καθεστώς της γλώσσας. Μια επίσημη γλώσσα της Ένωσης, τα Ιρλανδικά, ε, δεν μπορεί να μην έχει μέλλον. Είναι ένα πρόβλημα βασικό που μπορεί να, εξελιχθεί. Αν σήμερα δεν μπορούμε να παράσχουμε τα οικονομικά, πολιτικά και διοικητικά μέσα για να μπορέσουν να διατηρηθούν ε, οι γλώσσες. Γλώσσες που σήμερα δεν κινδυνεύουν μπορεί να κινδυνεύσουν. Τα εσθονικά, επίσημη γλώσσα της Ένωσης και τα γερμανικά κάποια στιγμή, γιατί όχι. Πρόκειται για μια διαβολική μηχανή, μηχανή της ενοποίησης, της εξομοίωσης του ομοιόμορφου, που είναι το αντίστροφο αυτού που θέλει η Ευρώπη. Η οικονομική λογική, η παγκοσμιοποίηση, οδηγεί όχι μόνο σε εξαφάνιση των γλωσσών, αλλά και σε μείωση του οικονομικού ιστού, άρα εις βάρος, εν τέλει, και ο σικολόγος το λέω αυτό, ε, εις βάρος της, οικονομικής, της ανάπτυξης η διαβολική αυτή μηχανή οδηγεί τα πάντα στα αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα φτωχαίνει όλες τις γλώσσες, τα γαλλικά, τα γερμανικά, και θα δημιουργήσει εν τέλει μια κουλτούρα χωρίς δημιουργικότητα. Και η δημιουργικότητα είναι που γεννά πλούτο, όχι το ομοιόμορφο. Είναι ένα βασικό ζήτημα και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τις σχετικές συζητήσεις ε, στο διάλογο και στην επίγνωση μπορεί και να μπορούμε να προχωρήσουμε ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η σατανική μηχανή. Ε, είναι δυνατό, γι' αυτό είπα, έδωσα το παράδειγμα της γλώσσας των Σάμι στη Φιλανδία, της Βασκικής στην Ισπανία. Η κατάσταση πριν από χρόνια ήταν χειρότερη από ό,τι είναι τώρα. Άρα η δράση δίνει αποτελέσματα και αυτό πρέπει να το έχουμε επίγνωση όλοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που καταγράφουν τον αριθμό των ομιλητών, των γλωσσών. Έχουμε στατιστικά για τη μείωση της απασχόλησης. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα θέματα, την διδασκαλία των γλωσσών αυτών στο σχολείο. Εγώ προέρχομαι από τη νότια Γαλλία, στην περιοχή μου μιλά, μιλάνε καταλάνικα. Ε, δεν είναι επίσημη γλώσσα, αλλά το, τη μιλάνε ένα εκατομμύριο άνθρωποι. 8 ε, εκατομμύρια άνθρωποι, συγγνώμη. Υπάρχουν στοιχεία για να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης πριν προχωρήσουμε προς άλλα μέτρα. Υπάρχει από το 1996 και μετά η UNESCO κάνει ένα παγκόσμιο ευρετήριο γλωσσών και η πλειοψηφία των γλωσσών ε, δεν είναι η Ευρώπη μόνο, είναι η Ινδική υποήπειρος, η Αφρική κλπ. Η Ένωση επίσης ε, εμπλέκεται. Το πρόγραμμα της UNESCO απειλείται και αυτό το ίδιο το πρόγραμμα το μόνο διεθνές πρόγραμμα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο απειλείται, γιατί όπως ξέρετε η UNESCO έχει σοβαρά προβλήματα ε, προπολογισμού μετά από πολιτικές αποφάσεις που έλαβε για την Παλαιστίνη. Πολλά προγράμματα αμφισβητούνται εν γέννη. Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα αυτό προχώρησε χάρη στην συνεισφορά μίας και μόνη χώρας, μίας και μόνης χώρας, την που έδωσε τα λεφτά. Τώρα, επιστημονικά αυτό στέκει. Έχει καμία τριανταριά εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο που, που εξετάζει μια σειρά κριτηρίων. με ε, μεταβίβαση γενεών, αριθμό ομιλητών, ποσοστό ομιλητών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό ή με τον πληθυσμό του συνόλου της χώρας. Ε, υπάρχει δουλειά. Και στην Ευρώπη ίσως πριν αν δεν, αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση ευρωπαϊκή για αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία, θα παραμένουμε αδύναμοι βλέποντας απλά την εξαφάνιση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς που επαναλαμβάνω ότι δεν έχει μόνο συναισθηματικό χαρακτήρα αλλά περιλαμβάνει και οικονομικές διαστάσεις. Ο τουρισμός για παράδειγμα. Ο τουρισμός εξορισμού πηγαίνει Προ μια ανακάλυψη. Αν το μόνο που ανακαλύπτεις είναι το ίδιο πράγμα από όπου φεύγεις, ο, ο τουρισμός θέτεται επαμφιβόλο. Και υπάρχει και μια ολόκληρη δημιουργικότητα. Η γαλλική πολιτιστική παραγωγή ε, χρησιμοποιεί την οξυτανική, τον πανιόλ. Ε, κάθε μικρή κουλτούρα συμβάλλει στην γενική κουλτούρα σε όλες τις κουλτούρες. Ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά υπάρχουν αξιόπιστα αποτελέσματα που δείχνουν ότι μπορούμε με συγκεκριμένες βράσεις να ανατρέψουμε την δυναμική, να επαναφέρουμε τη γλώσσα στους νέους, να δημιουργήσουμε μια γλώσσα που είχε χαθεί από τους παππούδες να εκενθαρρύνουμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συζητήσουν το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Παγιαδέλη, σύντομα αν γίνεται. Τον κύριο Αλφόνση για ε, όσα μας είπε, μια, τίθεται με την πρωτοβουλία του αυτή ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά πρώτον στον αλφαβητισμό, δεύτερον στον, στη συρρήκνωση των ε, επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν παράλληλα με την διατήρηση των μειωνοτικών γλωσσών. Ένα ερώτημα που απευθύνεται όχι μόνο στον κύριο Αλφόνση αλλά και στην Επιτροπή. Υπάρχει κίνδυνος η υποστήριξη των μειωνοτικών γλωσσών πέρα από την πολύ σημαντική ε, πολιτιστική ε, και πολιτιστική κυρίως περιουσία που καταθέτει ε, στην πολυμορφία της Ευρώπης να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο πολιτικό για αυτονομιστικές δράσεις. Αυτό είναι η μόνη αγωνία που έχω σε σχέση με τη διατήρηση της ε, γλωσσικής, ε, όχι διατήρηση, με τη διαφύλαξη των μειονοτικών γλωσσών σε επίπεδο πολιτικό. Και θα περίμενα μια απάντηση από τον κύριο Αλφόνση. Ευχαριστώ πολύ. Το πολιτικό θέμα είναι πάντα παρόν. Η απουσία απάντησης στο αίτημα των ενδιαφερομένων κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση στην διόνυση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα, όχι το αντίστροφο. Όσο περισσότερο η Ευρώπη και οι τοπικές δομές μπορούν να απαντήσουν στις ενδιαφερόμενες κοινότητες, σε περιφέρειες, σε δήμους, σε νομούς, διάφορα επίπεδα είναι, οργανωμένε διασυνοριακές μερικέ φορέ δομέ. Κάθε φορά που θα δίνουμε τη δυνατότητα στις κοινότητες αυτές να έχουν κάποιες πολιτικές που θα διασφαλίσουν την κουλτούρα και τη γλώσσα τους, μειώνουμε τα πολιτικά προβλήματα, δεν τα αυξάνουμε. thank you. Um, now, um, just to let you... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Φρονσού Αλφονσί θα παρουσιάσει την um, έκθεση του τον Απρίλιο και θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διαταξής μας, ε, που είναι το υπαριθμόν 7, η ανταλλαγή απόψεων με την ε, Σέτε Σόης Σέτε Λούνας, Λούας, συγγνώμη, ε, δεν ξέρω αν το προφέρω, προφέρω σωστά, λέει η Πρόεδρος, Στι 29 Μαου αποφάσισαν οι συντονιστέ να καλέσουν εκπροσώπους του φεστιβάλ αυτού για να κάνουν μια παρουσίαση στο, στην Επιτροπή μας. Το φεστιβάλ άρχισε το 1973 ε, με ε, εκπροσώπους ε, από χώρες εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βραζιλία, Ισραήλ, Μαρόκο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία και σκοπό έχει να προωθήσει την κινητικότητα των ε, δημιουργών και των ε, έργων τους, ε, όπως επίσης και την πολιτιστική δικυλομορφία και τον πολιτιστικό τουρισμό. Έχουν συμπεριλάβει τον Χωσέ ε, Σαραμάγκο, τον Πορτογάλο λομπελίστα ε, που πήρε τον Νομπέλ το 1998 και τον Άριο Φου ε, που πήρε τον Νομπέλ το 1998. Λάβαμε το πρόγραμμά του, ε, του φεστιβάλ αυτού. Σήμερα ε, υποδεχόμαστε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών από το φεστιβάλ. Δέκα εξ αυτών θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε μόνο μία ώρα για το θέμα αυτό, οπότε θα πρέπει να είστε σύντομοι. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Αμοντάνσα, για πέντε λεπτά και μετά οι υπόλοιποι θα πρέπει να ε, περιοριστούν ε, σε δύο λεπτά το πολύ. Δίνω λοιπόν πρώτα το λόγο στον διευθύντη του φεστιβάλ. Έχετε το λόγο. Buongiorno, ε, molte grazie. Καλημέρα και ευχαριστώ την Επιτροπή Πολιτισμού για αυτή την πρόσκληση. το φεστιβάλ Σέτε Σόι Σέτε Λούας των, ε, της μουσικής ε, κουλτούρας του μεσογειακού και πορτογαλόφωνου κόσμου γίνεται εδώ και 20 χρόνια πλέον σε 30 πόλεις από 11 χώρες που ανέφερε η πρόεδρος. Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία, Μαρόκο, Ισραήλ, Πράσινο Κροτήριο και Βραζιλία είναι το φεστιβάλ της κινητικότητας των καλλιτεχνικών έργων, των καλλιτεχνών και των θεατών από τον κόσμο της, τον πορτογαλόφωνο και μεσογειακό κόσμο. Έχει πρόεδρο, είχε πρόεδρο τον κύριο Ζωζέ Σαραμάγκο για 18 χρόνια, τον ε, Ντάριο Φώ και τώρα ο τελευταίος επίτιμος πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του Πράσινου Οκροτεδίου. Ο τίτλος ε, προέρχεται από το μυθιστόρημα του Σαραμάγκο. Ο Σαραμάγκο μας βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημα αυτού του φιλοδοξού έργου. Είναι το φεστιβάλ του υπτάμενου αυτοκινήτου που δημιουργήθηκε, της Πασαρόλα που δημιουργήθηκε το 1709 που στο μεμοριάλ του κομβέντου αναφέρει και ο Σαραμάγκο. Αυτή η πασαρόλα είναι το, το, σύμβολο του φεστιβάλ, το σύμβολο του διαφωτισμού και της ε, ανάδειξης ε, του ανθρώπινου πνεύματος. Γιορτάζει τη λαϊκή μουσική κουλτούρα. Είναι ένα φεστιβάλ με τρία πολιτισμικά κέντρα στην Ποντεβέρντα, στην Τοσκάνη, στην Πόντε Σόλ και στο Φροντινιάν, στην Νότια Γαλλία. Τα τρία αυτά κέντρα σε τεσσορίς προωθούν την, ε, την, ε, την ε, ανάδειξη των πλαστικών ατών, των πλαστικών συγγνώμη, τεχνών. Είναι το φεστιβάλ του Φάντο, του, του ρεμπέτικου, του φλαμένκου, της ευαρδίτικης μουσικής, των χοροδιών, των λαϊκών μουσικών της Νότιας Ιταλίας, της Βασκικής, της Οξυτανικής, της Βαλεντσιάνικης, της Ιστριακής μουσικής. Μουσικές που επανεξετάζονται από την σύγχρονη οπτική γωνία είναι το φεστιβάλ της παγκόσμιας μουσικής, της πορτογαλόφωνης και μεσογειακής μουσικής, το φεστιβάλ της διαφοροποίησης του μεσογειακού κόσμου, της διαφορετικότητας του μεσογειακού κόσμου και το φεστιβάλ που γιορτάζει τα σημεία επαφής μεταξύ των διαφόρων μουσικών ε, πολιτισμών του Μάρεν Όστρουμ. Είναι λοιπόν και το φεστιβάλ της παραγωγής πρωτότυπων μουσικών έργων πραγματικών ουσιαστικών ορχιστρών που συναθρίζουν νέες μουσικές, νέους μουσικούς από διάφορες χώρες της Μεσογείου που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά που μαζί παρέχουν, παράγουν ένα νέο ρεπερτόριο με βάση τις επιμέρους πολιτιστικές μουσικές κουλτούρες. Έχει πρωτότυπα χαρακτηριστικά και στις 30 πόλεις όπου λειτουργεί με, τον ίδιο, με το ίδιο όνομα προς τιμήν του Σαραμάγκου και την ίδια φιλοσοφία του προγραμματισμού. Θέλουμε να, να προγραμματίζουμε Πορτογάλους Ιτα, καλλιτέχνες στην Ιταλία, Ιταλούς στη Γαλλία, Γάλλους στην Κροατία. Ούτω ώστε το κοινό να εκτιμήσει και να γνωρίσει τον τεράστιο πλούτο της του πολιτισμού της Νότιας Ευρώπης. Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο μετήχαν άτομα όπως ο Σαραμάγκο, ο Φω, ο Κουστουρίτσα, η Ντούλσε Πόντε, η Μαρίζα Παρέδε, ο Νικόλα Πιοβάνι, ο Μανουέλ Ολιβέρη, η Λάουρα Μοράντε, ο Ζων Τζουγκιόνο Μπενάτο, η Τερέζα Σαλγκέρι, μεγάλε φωνέ του Φλαμένκο, Τενόρι, θα μιλήσει και εδώ, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι σημαντικό να φέρουμε εδώ την φωνή των καλλιτεχνών του φεστιβάλ. Κλείνω με την ελπίδα ότι η ουτοπιστική πτήση της Πασαρόλα αυτού του υπτάμενου αυτοκινήτου του Σαραμάγκο θα επιτρέψει να ενισχυθεί το αίσθημα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρίνο Μπουντίτσιν, αντιπρόεδρο της ε, τοπικού δήμου της, ε, στην Κροατία. Σας χαιρετίζω από την πόλη του Ροβίνιο και από την περιφέρεια της Ήμπριαν, μία από τις περιφέρειες της Κροατίας. Το Ροβίνιο είναι μία από τις έδρες του φεστιβάλ και αυτό δείχνει τον μεσογειακό μικρό κόσμο. Η περιοχή της Ίστρια, όπου βρίσκεται το Ροβίνιο, ήταν πάντα μια σημαντική περιοχή σύνδεσης της λεκάνης της Μεσογείου και του υποαλπικού και του κεντροευρωπαϊκού κόσμου. Οι βασικές αρμοδιότητες και ευθύνες του φεστιβάλ μας βρήκαν λοιπόν γόνιμο εξ αρχής έδαφος στην Ίστρια και στο Ροβίνιο που με το, με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την πολυεθνική, πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική ε, ταυτότητά της εκπροσωπεί όλες τις κουλτούρες της Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό και οι συμπολίτες μας και οι πάμπολοι τουρίστες που μας επισκέπτονται σε όλο το χρόνο θεωρούν το φεστιβάλ ως ε, στοιχείο κουλτούρας της Μεσογείου και εθνομουσικού πολιτισμού. Το φεστιβάλ, χάρη στο, στην οικουμενική γλώσσα που χρησιμοποιεί, τη μουσική δηλαδή, είναι ένα μοναδικό και ειδικό παράδειγμα της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του πολιτισμικού τουρισμού και των σημαντικών ευκαιριών για να γίνει γνωστή εκτός Ιστρίας και εκτός Κροατίας, για να γίνουν γνωστοί εκτός Ιστρίας και Κροατίας οι μεγάλες φωνές της μουσικής, της τοπικής και παραδοσιακής μουσικής. Ξέρετε ότι η Κροατία ετοιμάζεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να δούμε και την πρόκληση του συγκεκριμένου τομέα της προστασίας και της ανάδειξης της ε, πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τελειώνω. Η σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής υποστήριξης για τέτοια έργα είναι καθοριστική σημασίας. Είναι απαραίτητη ιδίω αν λάβουμε υπόψη τα τεράστια προβλήματα, ιδίω οικονομικού χαρακτήρα, που κατατρέχουν μια δημοκρατία όπως είναι η Κροατία, νέα δημοκρατία και που εξ αρχής θεωρεί ότι η είσοδος στην Ένωση και η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τους βασικούς δρόμους της μελλοντικής της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Κροατίας. Τώρα πάμε στον Αντώνιο Κάου από την Ιταλία. Io rappresento Από τη Σαρδινία πιο συγκεκριμένα. Καλημέρα σας. Νησί στο κέντρο της Μεσογείου είναι η Σαρδινία. Άρα, επειδή είναι στο κέντρο της Μεσογείου, είναι φυσικό να είναι σε ένα τέτοιο φεστιβάλ όπως αυτό που είσαι ο διευθυντή μας. Είναι νησί γεωγραφικά, αλλά και γλωσσικό νησί. Και μέσα στο νησί, σε αυτό το γλωσσικό νησί, υπάρχει και ένα πολιτισμικό νησί, που είναι η πολυφωνική χοροδία καν το ατενόρετο λέμε και το προστατεύει η UNESCO από το 2005 ως ε, κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτό το χοροδιακό είναι η παλαιότερη πολυφωνική χοροδία στον κόσμο, μοναδική στο είδος της και εμείς ε, ε, καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό αυτό το φεστιβάλ που μας αναδεικνύει γιατί ακριβώς αποτελεί μια ιδιαίτερη πραγματικότητα και δεύτερον διότι αισθανόμαστε σύγχρονοι στο μέτρο που περνούμε με τα τραγούδια και τα λόγια μας θεματικές της επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω με φωνικό τρόπο, με ωμέγα το φωνικό, ε, δύο-τρία τραγούδια μεταξύ φίλων. Αν μας το επιτρέπετε, θα σας τραγουδήσουμε αυτή την, με αυτή την πολυφωνία που νομίζω ότι δεν έχετε την ευκαιρία να ακούσετε κάθε μέρα. Αν συμφωνείτε, ελάτε εδώ, παιδιά. Βεβαίω, τραγουδίστε μας.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 Eh, Αυτές ε, οι πολιτιστικές ε, φωνές ε, που αποτελούν την έκφραση ενός ταβιστικού αρχαίγονου κόσμου θα θέλαμε να το τραγουδήσουμε περισσότερο, να τραγουδιέται περισσότερο και να μας επιτρέψει η παγκοσμιοποίηση και με τα εθνικά και διεθνή κονδύλια να μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της έκφρασης που πρέπει να προστατευτεί. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ όχι μόνο που μας μιλήσατε αλλά και που μας τραγουδήσατε. Πάμε τώρα στην Ελιζαμπέτα Ουντιβέρα από την Πορτογαλία. Σωστά λέω το, όνομά σας, παρακαλώ. Julgo Ε, και η πόλη μου αλλά και άλλες ε, πόλεις συμμετέχουν στο φεστιβάλ ε, Σέτε Σόης Σέτε Λούας. Παίρνουμε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις. Οι κοινότητές μας πρέπει να υποστηρίζουν τον πολιτισμό στην περιοχή μας το φεστιβάλ είναι πολύ κλασικό κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Πάντα λαμβάνει χώρα. Οι εκδηλώσεις πάντα ε, είναι, έχουν ε, όλα τους τα εισιτήρια ε, πουλημένα. Δεν βρίσκει κανείς θέση. Είναι πολύ δημοφιλές λοιπόν αυτό το φεστιβάλ. Και είναι και λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα όσα βλέπει κανείς στην τηλεόραση ή ακούει στο ραδιόφωνο. Βέβαια το 2013 θα είναι δύσκολο για όλους ε, γιατί δεν θα πρέπει να μειώσουμε μόνο τα, στον πολιτισμό τα κονδύλια αλλά και στην περιοχή μας το φεστιβάλ αυτό όντως θα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά το φεστιβάλ αυτό δίνει ε, χαρά, δίνει ελπίδα σε όλους του συμμετέχοντε, είναι ένα πολιτιστικό δίκτυο βοηθά όλους να δημιουργήσουμε, να υποστηρίξουμε μια πολιτιστική πολιτική, να, αλλάξουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να έρθουν νέοι από άλλες χώρες που θέλουν να πάρουν μέρος, να, να τους γνωρίσει ο κόσμος. Και το δίκτυο αυτό επιτρέπει την ε, ε, ανταλλαγή πληθυσμών, ε, καλλιτεχνών, μπορούμε να μάθουμε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και από τις υπόλοιπες βεβαίως πόλεις και χώρες που παίρνουν μέρος, να διδαχθούμε. Με την εκπόνηση του προγράμματος μας πάντα προσπαθούσαμε να διαφυλάξουμε και την ηλική και την άειλη κληρονομιά και για να είμαστε αποτελεσματικοί προσπαθήσαμε όλες αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Κλείνοντας να πω πολύ σύντομα ότι είμαι πολύ ε, ευτυχής που είμαστε σήμερα εδώ και παίρνουμε μέρος σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ζητήσουμε και εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες και εκπρόσωποι όμως της Περιφέρειας Νοήρας να κάνετε κι εσείς ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε τέτοιου είδους φεστιβάλ να συνεχίσουν να υπάρχουν για να συνεχίσουν να ενισχύουν την ε, ευρωπαϊκή πολιτιστική κουλτούρα. Αγαπούμε αυτό που γνωρίζουμε, λέει ένα παλιό ρητό. Ε, Όποιο λοιπόν δεν μα ξέρει, δεν ξέρει την περιοχή μα, καλό θα ήταν να έρθει γιατί θα την αγαπήσει σίγουρα. And now... Ευχαριστώ. Πάμε τώρα. Ε, κάποια εκπρόσωπος λείπει. Πάμε τώρα στον Χουάν Πινέγια. Εκπροσωπεί την Ισπανία. Ε, buenos días a todos. Καλημέρα σας. Εγώ εκπροσωπώ το φλαμένκο, τραγουδάω φλαμένκο, είμαι κανταόρο και τη μουσική της Νότιας Ισπανίας λαϊκής προέλευσης από έναν λαό που ήταν περιορισμένος, στερημένος της ελευθερίας αποτέλεσμα αυτής της ε, ανάγκη έκφραση ήταν το φραμένκο, το πιο γνωστό ε, το πιο γνωστό μουσικό έργο της Νότιας Ισπανίας και που ορίστηκε πριν από ένα χρόνο και σαν κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO. Αυτό, αυτή η επίσημοποίηση έδειξε κάτι το αυτονόητο, ότι είναι οικουμενικό το φλαμένκο. Το φλαμένκο, όπως κάθε κουλτούρα, υποφέρει από τις επιπτώσεις της κρίσης και της δημοσιονομικής κρίσης και θέλω να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα του φεστιβάλ σε Τεσόη, σε τη δυνατότητα διεξαγωγής αυτού του φεστιβάλ, ώστε μια τόσο σημαντική μουσική όπως το φλαμένκο να φτάνει στα πιο κρυφά σημεία της Ευρώπης. Όχι κρυφά, αλλά σε σημεία όπου ε, ήταν δύσκολο να φτάσει η μουσική αυτή αυτό είναι το βασικό μεγαλείο του φεστιβάλ για μένα. Είναι σημαντικό σε αυτή την πολιτισμική συνάντηση να είμαι παρόν και να παρέχουμε τα στοιχεία που ζητάτε. Να είναι μια, δουλειά, μια δουλειά όπου η παραδοσιακή μουσική, το φλαμένκο από την Αμανταλουσία, οι ιταλικές, οι κροατικές, οι πορτογαλικές μουσικές, η μουσική από το Ισραήλ να συμμερίζονται το ίδιο έργο και να πλουτίζουν η μία από την άλλη. Βουάντε Ετεσόης, η φωνή της Ετεσόης είναι μία συνύπαρξη όχι μόνο μουσικής που είναι σημαντική αλλά και μιλώ και με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Αφλόνση επαναφέρει και μία γλώσσα που μιλιόταν παλιότερα στη Μεσόγειο και που λέγεται Σαμπίρ. Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα αυτή για να μιλούμε όλοι μαζί βάση, πάνω στο Σαμπίρ. Η συνύπαρξη αυτή που δημιουργεί το φεστιβάλ είναι ήδη εξορισμού κάτι σημαντικό για την ε, συνύπαρξη, τιμή θρησκευτική συνύπαρξη. ένα Ισραηλινός τραγουδιστής, ένα μουσουλμάνο ή ένα χριστιανό μουσικό, άθεοι που συνυπάρχουν βάσει τη μουσική και προωθούν τον πολιτισμό. Να σας ευχαριστήσω εκ νέου που μου δώσετε το λόγο να μιλήσω και να σας ζητήσω να αγωνιστείτε ούτως ώστε οι πολιτικουλτούρες μην... Εγώ είμαι από τη Γρανάδα, εκεί που γεννήθηκε ο Λόρκος συμπολίτη μου και έλεγε ότι αν ένα άτομο πεινά μην του δώσεις μόνο ψωμί αλλά ψωμί και ένα βιβλίο διότι με το βιβλίο, με τον πολιτισμό θα μάθαινε να κερδίζει το ψωμί του. Ζητώ λοιπόν να βοηθήσετε για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το ΣΕΤΕ ΣΟΙ ΣΕΤΕ ε, σε και τελειώνοντα θα μου επιτρέψετε να σας τραγουδήσω ένα φλαμένκο πρωί. Ξέρετε εμείς το φλαμένκο νύχτα το τραγουδάμε συνήθως αλλά αν μου επιτρέπετε να σας τραγουδήσω ένα φαντάγκο.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 Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που συνδέσατε και τούτο το σημείο της ημερήσιας διάταξης με το προηγούμενο, την έκθεση δηλαδή του κυρίου Αλφόνση. Προχωρούμε με την κυρία Πιλάρ Αλτοτάλενς, πάλι πρόσωπο της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνει η Επιτροπή Πολιτισμού του Κοινοβουλίου για να σας μιλήσουμε για το πολιτιστικό δίκτυο ΣΕΤΕΣΟΙΣ Τα Η... Ταβέρες Δεβαϊδίνα είναι μια παράκτια πόλη με 18.000 κατοίκους νότια της Βαλένθια. Από το 1997 το Ταβέρνες έγινε η έδρα στην Ισπανία του ΣΕΤΕΣΟΙ Ετελούες. Λάβαμε προ, μουσικές προτάσεις, καλλιτεχνικές προτάσεις και θεατρικές προτάσεις από τις διάφορες χώρες που μετέχουν στο φεστιβάλ και κάναμε και οργανώσαμε και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης επιτρέψαμε σε θεατρικές και μουσικές ομάδες της Βαλένθια να παίξουν μέσα στο πλαίσιο του ΣΕΤΕΣΟ ή ΣΕΤΕΛΟΑΣ. τη συμμετοχή στο κοινοτικό έργο συνεργασίας πολιτισμικού χαρακτήρα του 2005 Interreg 3, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο έργο ε, πολιτιστικού χαρακτήρα που υποστηρίζει ο Δήμος μας συνεχώς. Είμαι βέβαιη ότι χωρίς την κοινοτική υποστήριξη και χωρίς το δίκτυο σε σε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πλούτο που δημιούργησαν οι δυναμικές των αλλαγών και που συνεχίζουν να δημιουργούν. Η σπουδαιότητα της τοπικής, ε, των τοπικών αρχών είναι όλο ένα και μεγαλύτερη. Οι πόλεις αποκτούν βασικό πρωταγωνιστικό χαρακτήρα. Η συνεργασία αποκτά έτσι μεγαλύτερη αξία και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ενίσχυσης του τοπικού ρόλου ως υπεύθυνο ε, για τη, το, τον πολιτισμό ε, στο Δήμο θέλω να υπογραμμίσω ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ούτω ώστε και εκπαιδευτέ και εκπαιδευόμενοι να μάθουν καλύτερα την πολιτιστική τους, ε, τον πολιτικό του πλούτο και να ενισχύσουν την δηλαδή αυτή μέσω διαφόρων δομών που επιτρέπουν τον διάλογο και που μετατρέπουν τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους σε υποκείμενα. Ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, τα βιβλία δεν είναι μόνο υλικό εργαλείο, ιδίω αυτή τη δύσκολη εποχή είναι αναγκαία εργαλεία για να αναπτυχθούν. Γι' αυτό σας ζητώ να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε νέους δρόμους μέσω του διεθνούς, του διεθνούς δικτύου σε Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε μια κυρία από τη Γαλλία τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχάς ε, την Επιτροπή σας που μας δίνετε τη δυνατότητα να παραστούμε εδώ σήμερα σε σχέση με την εμπειρία μας ε, στο φεστιβάλ ε, αυτό. Είμαι από το Φροντιλιέ, 23.000 κάτοικοι στην Νότια Γαλλία, στη Μεσόγειο, στο Λονγκτό Κρουζιγιόν. Ε, είναι ανάμεσα στον ορεινό όγκο και στη Μεσόγειο και μάλιστα ε, είναι ο παραγωγός περιοχή. Ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε περήφανες γυναίκες από την, για την καταγωγή τους. Υπάρχουν επίσης πολλοί Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι και Μαροκινοί μετανάστες ε, είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται να συναντήσουμε άλλους δημιουργείς, το, δημόσιο, το, το, το, κοινό, ε, μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε την παραγωγή μας, ε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας καταλάβουν καλύτερα την κοινωνία μας, να διαδώσουμε την, τα, την καλλιτεχνική μας παραγωγή και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Γι' αυτό ακριβώς ε, μας δίνει τη δυνατότητα το φεστιβάλ αυτό να παρουσιάζουμε Ευρωπαίους ε, δημιουργούς αλλά και τοπικούς ε, δημιουργούς, τοπικούς καλλιτέχνες και στις πλαστικές τέχνες και στη μουσική. Κάθε καλοκαίρι έχουμε ένα τεράστιο ραντεβού που είναι το αποκορύφωμα των προσπαθειών μας όλης της χρονιάς και από το 2010 έχουμε και ένα κέντρο σε Τελούα. Ε, για να προωθήσουμε την περιοχή της Μεσογείου ε, με την εκπροσώπηση όλων των δημιουργών από τις περιοχές τους ώστε να μπορούν να ε, κινηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τοπικοί μας καλλιτέχνες. Επίσης προσπαθούμε να αγγίξουμε τους νέους και τους επισκέπτες μας στο, με όλους τους ε, υπόλοιπους καλλιτέχνες μπορούμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου ε, και ε, λόγω της υποδοχής τους στο φεστιβάλ αλλά και λόγω της γνωστοποίησης της καλλιτεχνικής μας παραγωγής μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να γνωστοποιήσουμε την πολιτιστική μας παραγωγή και να ενθαρρύνουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ραούλ Ταμπέρα Πίντο από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, είμαστε εδώ και 17 χρόνια στο φεστιβάλ αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ με χαρακτηριστικά ε, εντελώς ε, μοναδικά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν οι νότιες χώρες που τόσο πολύ επικρίνονται ανέλαβαν πρωτοβουλίες ε, σε πολιτιστικό επίπεδο και είναι έτσι ε, πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ένα τόσο μοναδικό φεστιβάλ ε, στην Ευρώπη που αφορά την Μεσόγειο που είναι το λίκνο το πολιτιστικό της Ευρώπης ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την περιοχή αυτή με θετικότερο τρόπο. Οι τοπικές αρχές ε, παρεμβαίνουν με αποτελεσματικό τρόπο ώστε αυτό το φεστιβάλ ε, να μπορεί να λάβει χώρα. Επίσης, η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει τη σημασία αυτών των φεστιβάλ. Εκτός από την προώθηση των ε, καλλιτεχνών, κάνει πολύ περισσότερα μέσω των εργαστηρίων ε, καλλιτεχνών, ε, στους οποίους δίνεται έτσι δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες, ε, με ηθοποιούς δηλαδή, με ζωγράφους και... και τους δίνει τη δυνατότητα να αγγίξουν περισσότερο θεατές που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να ε, αγγίξουν. Είναι λοιπόν πολύ μοναδικά τα χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας. Όλες οι πόλεις που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι πάρα πολύ σημαντικές. γνωστοποιούμε και άλλα πράγματα, την ε, γαστρονομία και το καλό κρασί της Μεσογείου. Τόνι Ρέλη, from Italy. από την Ιταλία. Ευχαριστώ. Πρώτον, ε, σας ευχαριστώ πρόεδρε και όλα τα μέλη που μας δώσατε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε το έργο σε τεσόης τελούας. Όπως είπατε το έργο γεννήθηκε το 1993 στην Ποντεβέρα την πόλη που εκπροσωπώ σήμερα το πρωί από μια ομάδα νέων πτυχιούχων μεταξύ των οποίων ο κύριος Μποντα, ο Μάρκο Μποντάντσα ο οποίο ήθελε να γνώσει με πιο βαθύ τρόπο την πολιτιστική κουλτούρα της Μεσογείου. Ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ αυτό ήταν ότι ε, η... δεν ήταν μόνο γνώση της μουσικής, αλλά παρουσίαση των βασικών, των καλύτερων καλλιτεχνών της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Νότου. Μέσω των ανταλλαγών αυτών περνάει η παράσταση πέρα από τη χώρα της προελευσής και επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίσουν πολιτιστική πραγματικότητα άλλων χωρών. Πιστεύω ότι επιτρέπει σε εκείνους που για οικονομικούς λόγους ίσως δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό να καλύψουν το πολιτιστικό κενό μεταξύ των πολιτών. Αυτό ισχύει για τη δική μου πόλη, αλλά ισχύει και για τις άλλες πόλεις του, που, όπου είναι το φεστιβάλ, που απέκτησε ένα κοινό που ξεπερνά το έδαφος τη συγκεκριμένη περιοχής. Τα τελευταία χρόνια η εμπειρία πλούτησε με τη δημιουργία τριών κέντρων, ιδίων στην Ποντεντέρα, άνοιξε το 2009 ε, ένα τέτοιο κέντρο το οποίο χρησιμοποίησε την τοπική ε, παραγωγή της, την, την υποστήριξη της Πιάτζιο που φτιάχνει την Βέσπα και που ε, είναι στο κέντρο της παραγωγής στην ε, περιοχή μας. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτισμικών γνώσεων μεταξύ περιοχών και, και ε, πολιτών και επέτρεψε την διεύρυνση του φεστιβάλ και σε άλλους τομείς της τέχνης, τη σύγχρονη τέχνη για παράδειγμα. Έτσι έχουμε εκθέσεις, παρουσίαση βιβλίου και έκθεση ε, και εκθέσεις τέχνης παιδιών. Να υπογραμμίσω ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική στιγμή ο συντονισμένος προγραμματισμός και μουσικά και από την άποψη της σύγχρονης τέχνης επιτρέπει να γίνουν οι δραστηριότητες αυτές με περιορισμένο κόστος. Εν τέλει, όπως τα τελευταία χρόνια ε, η ανταλλαγή των στοιχείων αυτών είναι ένα μέσο για να, γίνει γνωσ... για να γίνουν γνωστά η παραγω... για να γίνει γνωστή η παραγωγή όλων των πόλων και ιδίως την παραγωγή της δικής μας πόλης σε άλλες. Ευχαριστώ. Έχουμε μια εταιρεία παρέμφαση του Αγκούστο ε, Μιλάνα. Ωραία, έχετε το λόγο και είστε ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ήθελα να μιλήσω από μια διαφορετική εμπειρία, την εμπειρία μιας μικρής, ενός μικρού χωριού νότια της Ρώμης που έχει μια ένα πολιτιστικό πλούτο. Είχαμε στη δεκαετία του 50 καλλιτέχνες εθνικής εμβέλειας στην ε, ζωγραφική στο Τζεζεντσάνο με μια ιστορική ε, παρουσία αλλά όταν έγινα υπεύθυνο ε, πολιτισμού στο Δήμο διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε σύνδεση αυτής της, του τοπικού πλούτου με τον πλούτο άλλων χωρών. Η εμπειρία μου λοιπόν ερχόταν από την, το, το, το διεθνές πλαίσιο. Δούλευα στη δεκαετία του 70 στις Βρυξέλλες και είχα ασχοληθεί ε, με την ε, επέκταση του πολιτισμού στην Ευρώπη. Το φεστιβάλ αυτό ήταν η ευκαιρία για να μπούμε στο δίκτυο αυτό με μεγάλες ε, της διοίκησης των διοικήσεων και το φεστιβάλ αυτό γίνεται στο Τζεζεντσάνο εδώ και τα τελευταία χρόνια με χαρακτηριστικά που ήδη υπογραμμίστηκαν για πρώτη φορά σε, μια, σε ένα χωριό 40 χιλιόμετρα από τη Λόμη ακούστηκε για πρώτη φορά το πορτογαλικό φάγκντο μουσική από το Ισραήλ από περιοχές της Μεσογείου που ουδέποτε θα είχαν ε, φτάσει στα αυτιά μας, διότι η μουσική αυτή είναι τοπικού χαρακτήρα. Και πρέπει να τονίσω ότι είναι δύσκολο σε έναν υπεύθυνο πολιτισμού να περάσει αυτή την άποψη σε τοπικό επίπεδο. Να καταλάβει δηλαδή ότι είναι καλύτερα να έχουμε τρεις μέρες διεθνές φεστιβάλ παρά να έχουμε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις ε, τοπικού χαρακτήρα. δημιουργήσαμε αυτό το φεστιβάλ όχι μόνο για να γνωρίσουμε την μουσική των άλλων περιοχών, αλλά για να ενισχύσουμε και την τοπική εμπειρία, την τοπική παραγωγή μουσικής. Γι' αυτό στο χωριό μου ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ε, ξανά την ε, μουσική των άλλων χωρών και δημιουργήσαμε μια ορχήστρα χρωμάτων που λειτουργεί είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ με, πάνω από μέχρι και 50 όργανα και, και έγχορδα και πνευστά με δικό της πρόγραμμα μουσικής όλης της Μεσογείου από όλους ε, τους χώρους. Έχουμε, έχουμε, υπάρχει μια ομάδα από την Ίστρια, οι οποίοι ήρθαν στο Παλκοσένικο και ε, στη σκηνή και έπαιξαν δικά τους κομμάτια. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί πλούτο, επαγγελματικό πλούτο νέων, που κατόπιν θα γίνουν η μουσική της, του αύριο. Και θα θεωρήσουν ότι η εμπειρία αυτή είναι πλούτος της προσωπικότητάς τους. Μια τελευταία παρατήρηση. Πόσο η σημαντική είναι η υποστήριξη της Ευρώπης. Το κατασκεύασμα που δημιουργήσαμε σε τοπικό επίπεδο για να διατηρηθεί το φεστιβάλ είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Χρειάζεται, χρειάζονται πόροι από την περιφέρεια, από τον νομό, χρειάζονται διαγωνισμοί, χρειάζονται αναθέσεις, περίπλοκες διαδικασίες που καθιστούν δύσκολη και προσωρινή την δημιουργία αυτού, την συνέχιση αυτού του έργου που απαιτεί ωστόσο μακροπρόθεσμη προοπτική. Γι' αυτό η υποστήριξη της Ευρώπης είναι σημαντική. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Thank you to all of you. Ευχαριστώ όλους. Ήταν πολύ καλή ιδέα να σας ε, ε, καλέσουμε εδώ, να ακούσουμε τις απόψεις σας, ε, να ε, μας πείτε να, τι ακριβώς κάνετε στο φεστιβάλ και βεβαίως να μας δείξετε πώς ακριβώς συνεργάζεστε και τι σημαίνει να έρχονται σε επαφή τόσοι ξεχωριστοί διαφορετικοί καλλιτέχνες από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς σημαίνει και βέβαια πάντα θέλουμε να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν ε, να πάρουν το λόγο και η Κομισιόν βεβαίως. And then Mrs. Costa. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους του Φεστιβάλ Σετεσόης Σετελούας. Ίσως να μην ξέρει κανείς ε, από πού προήλθε αυτό το όνομα του φεστιβάλ. Το όνομα αυτό είναι το, ο τίτλος ενός μυθιστορήματος ε, του Σαραμάγκου. Υπήρχαν δύο χαρακτήρες ε, μέσα στο ε, μυθιστόρημα που είχαν αυτά ακριβώς τα ονόματα. Ο ένας ζει το πρωί και ο άλλος ζει το βράδυ. Και φαίνονται στο μυθιστόρημα οι διαφορετικές ε, πτυχές της προσωπικότητας αυτών των δύο χαρακτήρων κανείς δεν βλέπει τα πάντα, κανείς ε, δεν ξέρει τα πάντα. Αυτό δείχνει το μυθιστόρημα, την διαφορετική οπτική γωνία των ε, ανθρώπων. Και αυτό που βλέπει κανείς το πρωί, ε, το βράδυ μπορεί να το δει με τελείως διαφορετικά μάτια. Έχουμε μια Ευρώπη που είναι χωρισμένη και αυτή στα δύο. Και Καμιά φορά λέγεται ότι η μεν είναι η καλή, η μεν είναι κακή, ο ένας είναι πιο δυνατός, ο άλλος είναι πιο αδύναμος στην Ευρώπη. δεν χρειάζονται τέτοιες ε, δηλώσεις βεβαίως, δεν βοηθούν να βγούμε από την ε, κρίση. Και ο πολιτισμός είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για να βγούμε από την κρίση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε βέβαια και την οικονομία αλλά και, την, ε, και τον πολιτισμό και πέρα από αυτό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μέσω του πολιτισμού και τις αρνητικές συνέπειες που έχει φέρει η κρίση σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό ε, να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για την ε, αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ε, δυνατότητες. Και ε, τα δύο αυτά, ε, τους δύο αυτούς τομείς παράνομης δραστηριότητες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε εφόσον θέλουμε να έχουμε δημοκρατικές κοινωνίες. Έχω ένα ερώτημα για την άλλη πλευρά της ε, Μεσογείου. Ε, μιλήσατε για το Ισραήλ. Με τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης τι γίνεται. Αυτές οι χώρες δεν θα πρέπει να συστρατευτούν στο, σε αυτό το φεστιβάλ. Μήπως πρέπει εμείς να τίνουμε μια χείρα ε, βοηθείας και στήριξης προς αυτούς γιατί είναι σημαντικέ και οι χώρες αυτές για την σταθερότητα όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και για τις ε, χώρες της ε, Νότιας Ευρώπης, τις περιφερειακές χώρες. Ε, πάντα σκεφτόμαστε ότι η Μεσόγειος είναι το όριο και μετά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως υπάρχουν και άλλες χώρες πέρα από τη Μεσόγειο και αν θέλουμε να έχουμε σχέσεις με, την, ε, με τις χώρες της Αφρικής, τότε αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα μέσω του πολιτισμού. Εκεί δεν χρειαζόμαστε ούτε διάσωση, ούτε πακέτα λιτότητας, ούτε τίποτα. Ε, τι είδους λοιπόν... Ε, συμμετοχή θα μπορούσε να υπάρξει ή τι είδους ε, νομική οδός θα χρειαζόταν έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος και αυτές οι χώρες και στο δικό σας αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά ε, φεστιβάλ που γίνονται. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον και σε σχέση με την Ειδική Επιτροπή για, την, για το Οργανωμένο Έγκλημα να το σκεφτούμε και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε τον πολιτισμό αλλά και τέτοια φεστιβάλ όπως οργανώνετε εσείς να τα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. θα μπορούσε ας πούμε, κανείς να πει ότι θα μπορούσαμε να δεσμεύσουμε τα χρήματα του οργανωμένου εγκλήματος και να, τα, να, να μπουν σε ένα ε, ε, ευρωπαϊκό ταμείο και μετά να δοθούν για ευρωπαϊκές πολιτιστικές δραστηριότητε. Οι πολίτες ε, θα πρέπει να να γνωρίζουν, να μπορούν να υποφεληθούν από αυτά τα, τα μαύρα χρήματα. Θα μπορούσε ίσως λοιπόν αυτό να αποτελέσει ένα κομμάτι της πολιτικής για τον ε, πολιτισμό. Και επίσης θέλω να πω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε και το πρόγραμμα Οδυσσέας το οποίο βασίζεται στην καινοτομία, στο διάλογο, ως λύσεις, ως ε, τρόπους ε, εξόδου από την κρίση. τρεις, τρία μεγάλα πνεύματα α, ενώθηκαν γι' αυτό. Ένας Άραβας φιλόσοφος, ένας Εβραίος φιλόσοφος και Προσπαθήσαμε με βάση και, την, και το πρόγραμμα που υπάρχει για τον διαπολιτισμικό διάλογο αλλά και για τον, με το θρησκευτικό διάλογο να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση που δεν ήταν μόνο ε, φωνη, ε, που, όπου η φωνητική ακρόαση είχε πολλές διαστάσεις. Η έρευνά σας ε, είναι πολύ σημαντική ε, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε για τις γλώσσες που κινδυνεύουν. Τώρα μιλάμε για τους ήχους που κινδυνεύουν στη Μεσόγειο και για τις νέες ε, μορφές ε, του, της μουσικής, το φλαμένκο που συνυπάρχουν στην εμπειρία αυτή. στη φάση αυτή θέλω να σας συγχαρώ για τα 20 χρόνια της εμπειρίας σας, πλούτησε ο χώρος σας με 25 πόλεις ε, που μετέχουν πολίτες, τοπικές αρχές ε, και όπου μαζί συνυπάρχουν πραγματικότητες που επιτρέπουν μια σημαντική ομαδική δουλειά. Προσωπικά είχα εμπλακεί στην ε, δραστηριότητά σας αυτή γιατί είμαι εισηγήτρια για την Δημιουργική Ευρώπη, ένα νέο πρόγραμμα της Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια για την πρόθεση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη. Το κάναμε και με την Επιτροπή ε, στο παρελθόν. Υποστηρίζουμε Υποστηρίζουμε την ε, παραγωγή στα φεστιβάλ και οπτικοστικά και πλαστικών τεχνών για την πρόθεση νέων έργων, την ε, συνύπαρξη παλιάς, πα, ε, και σύγχρονης μουσικής, κάτι που βεβαιώνει η δική σας εμπειρία. Κάτι άλλο που, με το οποίο συμφωνώ μαζί σας είναι το ότι ξαναφέρουμε στο κέντρο του ευρωμεσογειακού διαλόγου μέσω του πολιτισμού την μετατροπή της Μεσογείου σε ένα χώρο συνάντησης, όχι διαφωνίας. Κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη του σήμερα. Δύο ερωτήματα λοιπόν θέλω να θέσω. Πρώτον, μιλούσατε για τις δυσκολίες ε, Έρχομαι από την ίδια περιοχή μέσα στη Ρώμη. Τι δυσκολίες οικονομική υποστήριξη. Είχατε τα τελευταία χρόνια εξετάσει τις δυνατότητες που δίνουν τα διασυνοριακά ταμεία που είναι μια ευκαιρία για σας. Δεύτερο. είμαι η και στην Επιτροπή Γυναικών για την κατάσταση των γυναικών μετά την ε, Αραβική Άνοιξη. Μετέχουν εκεί, μετέχουμε σε ένα δίκτυο με γυναίκες βουλευτές της, Βορείου Μεσογείου, της Νότιας Μεσογείου. Ρωτώ, έχουμε διμερείς ε, συμφωνίες που ενισχύθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν με χώρες της Νότιας Μεσογείου που περιλαμβάνουν και διάσταση εκδημοκρατισμού. Εκεί περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των πολιτισμών. Το έχετε υπόψη σας, εμείς προτείναμε το θέμα της κυκλοφορίας των γυναικών, των γυναικών καλλιτεχνών, των γυναικών πολιτισμικών δημιουργούν να είναι ένα μέτρο υποστήριξης και το και τούτο παρέχει μεγαλύτερες ε, δυνατότητες για να υπάρξει υποστήριξη και για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει η κουλτούρα ένα μέσο συνάντησης και δημιουργίας. Κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί και δεν πρέπει να περικοπεί λόγω κρίση, γιατί αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον και για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σκούρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας, γιατί μας εξήγησαν και μας επέτρεψαν να ακούσουμε συνθετικά και σύντομα το πνεύμα που θα πρέπει να μας διέπει. Το απόγευμα θα συζητήσουμε με την Ιρλανδική Προεδρία για να καταλάβουμε τους στόχους της νέας Προεδρίας στον τομέα του, του πολιτισμού, της κουλτούρας. Πέραν των ε, μεγάλων στρατηγικών ε, που πρέπει να λάβουμε, η απάντηση είναι αυτή που ακούσαμε και αισθανθήκαμε σήμερα. Η ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων πρωτοβουλειών με ενθάρρυνση των ήδη φυστάμενων προγραμμάτων, ούτω ώστε να στηριχθεί η Ένωση στην εμπειρία αυτή κανονικά αυτή την ακρόαση δεν πρέπει να την κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά ίσως στην Οικονομική Επιτροπή. Την, ε, εκεί όπου θα μπορέσει ίσως να γίνει κατανοητό ότι οι επιλογές Ξέρουμε τι γίνεται αυτό τον καιρό με τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό αλλά ο στόχος θα πρέπει να είναι η Ευρώπη να μπορέσουμε να βρούμε νέους τρόπους υπέρβασης της κρίσης που δεν θα στηρίζονται μόνο σε οικονομικές παραμέτρους αλλά που θα έπρεπε να επιτρέπουν να καταλάβουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να βοηθήσει την επίλυση και άλλων ζητημάτων. Ο πολιτισμός, και αυτό το λέω ε, για, δεν θέλω να ενοχλήσω τον κύριο Μπαρόζο, αλλά νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν είναι θέμα μόνο της Επιτροπής Πολιτισμού. Εμείς θα πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Συμφωνώ με τα αιτήματα των συναδέλφων. Είναι ενδιαφέρον να καταλάβουμε και λειτουργικά ποια είναι τα μέσα που καλύτερα μπορούν να διατεθούν για, την, ε, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την εμπειρία αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Okay, now I would like to ask the Commission. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί. Α, δεν θέλει. Καλά. Εντάξει, τότε ο διευθυντή του φεστιβάλ να λάβει το λόγο. Θα τα πω στα πορτογαλικά. Για να σεβαστώ την ε, πολιτιστική ποικιλομορφία του φεστιβάλ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Το φεστιβάλ είναι υποψήφιο σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα χρηματοδοτηθεί ή όχι. Όπως και να έχει πάντως, ελπίζουμε οι χώρες ε, της ε, Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής εννοώ να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Στο πλαίσιο κάποιων προγραμμάτων ελπίζω να μπορούμε 15% των ε, του, προπολογισμού του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητές μας να τις ε, χρησιμοποιήσουμε, να, το χρησιμοποιήσουμε για ε, δραστηριότητες εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φεστιβάλ είχε ήδη παρουσία στο Ισραήλ και το Μαρόκο. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζει, να, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει ε, να μας υποστηρίζουν ε, οργανώσεις οι οποίες ε, στο παρελθόν μας υποστήριξαν στην προσπάθειά μας αυτή. Υπάρχει ένας διάσημος ζωγράφος μαροκινός σε μία πόλη στο Ισραήλ, ο οποίος ζει μάλλον λαθρέα στην περιοχή γιατί είχε προβλήματα θεωρήσεων και δεν ε, υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς τον προσκαλέσαμε τον ε, ζωγράφο αυτό ε, όταν είχαμε πάει στο Ισραήλ και σας το λέω απλώς για να σας πω τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε γιατί η νομοθεσία δεν προστατεύει τους καλλιτέχνες, η υφιστάμενη νομοθεσία. Έχουμε μάλιστα και μία πολυμερή ορχήστρα με μουσικούς από την Αλγερία, την Τινησία, και την Αγέμ, η οποία είναι μια πολύ γνωστή ε, τραγουδίστρια που ήταν η φωνή της ε, επανάστασης στην Τινησία. Αλλά αυτό βέβαια ε, κατέστη δυνατό μόνο και μόνο χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, για να σας ζητήσουμε να μας βοηθήσετε στην συνέχιση της προσπάθειάς μας αυτής και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρούσα εδώ σήμερα Εμείς υποβάλαμε την, την υποψηφιότητά μας για να μπορούμε να λάβουμε χρηματοδότηση. Ο κύριος Ταβάρης μίλησε για τη δυνατότητα διευκόλυνση θεωρήσεων για τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ. Αυτή είναι εξαιρετική ιδέα. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι γεγονός ότι στις χώρες που πηγαίνουμε δεν έχουμε καμία προστασία και μετακινούμεθα χωρίς καμία νομική πλαισίωση. Και καμιά φορά ε, η συμπεριφορά στους ε, καλλιτέχνες είναι πραγματικά πολύ ταπεινωτική κατά τις μετακινήσεις τους. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Το Ίδρυμα Αναλίντ μας βοηθά πολύ. Στην Τινησία θα ανοίξουμε ένα καινούριο κέντρο προκειμένου να έχουμε, παρουσία και εκεί, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια ώστε να υποστηριχθούμε και από τους δήμους και τις κοινότητες της, ε, του αραβικού κόσμου που δεν γνωρίζουν την ιδέα αυτής της ε, ενίσχυσης. Πρόκειται λοιπόν για μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση, μας ε, είπε πολλά πράγματα η ε, Σίλβια Κώστα, περιέγραψε πολύ σωστά την ε, κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να υποφεληθούμε από τις συμφωνίες αυτές για να εξελίξουμε τις προσπάθειές μας. Το άνοιγμα στην νότια ε, όχθη της ε, Μεσογείου θα έχει σημαντικό οικονομικό όφελος. Ε, είναι μεγάλες οι αγορές εκεί που είναι σημαντικές και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο. Ο πολιτισμός μπορεί έτσι να ανοίξει νέες αγορές στον αραβικό κόσμο. Από πλευράς αραβικού κόσμου τώρα υπάρχει κάποια θέληση να ε, γνωρίσει καλύτερα τον ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά είναι πολύ ε, κακώς οργανωμένη. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα σημαντικός συνομιλητής ε, στο πλαίσιο του, της λεκάνης της Μεσογείου. Έχουμε ένα δίκτυο που υποστηρίζει τους καλλιτέχνες αυτούς και είναι πολύ σημαντικό αυτό για σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, δεν θα ήταν δυνατόν να οργανώσουμε το φεστιβάλ χωρίς την υποστήριξη των καλλιτεχνών που πιστεύουν πραγματικά στην προσπάθεια αυτή. Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στην παρουσία του Ντάριο Φώ, του, ε, Ζωσέ, του Χωζέ Σαραμάγκο, που υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας και ελπίζουμε ότι οι σχέσεις με το Κοινοβούλιο και, και την Επιτροπή θα συνεχιστούν ώστε κάποια στιγμή σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία είτε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα να μην μας εγκαταλείψετε, να μην εγκαταλείψουμε αυτό το, την πολύτιμη κληρονομιά την οποία χτίσαμε εδώ και δύο δεκαετίες. Ελπίζουμε ότι το φεστιβάλ θα εξακολουθήσει να παραμένει ένα μεγάλο γεγονός κατέρωθεν ε, της Μεσογείου. Ελπίζουμε να παραμείνει μια πραγματικότητα και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο ενός διαλόγου μεταξύ διαφόρων πολιτισμών και ειδικότερο ε, μεταξύ των Ισραηλινών, των Αράβων και των υπολείπων της ε, λαών της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, ως ε, Επιτροπή πάντα προωθούμε έναν ε, φιλόδοξο προϋπολογισμό για τον για τον πολιτισμό. Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει μεγάλη αντίθεση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι χώρε που συνεισφέρουν θέλουν να τον μειώσουν. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε να αυξηθεί ο προπολογισμό για την εκπαίδευση και, την, και τον πολιτισμό. Αλλά ο κύριο ο κύριος Κάμερον και κάποιοι άλλοι αντιδρούν, κάποιοι άλλοι κρατών και κυβερνήσεων όπως θα ξέρετε, αντιδρούν. Οπότε δεν είναι εύκολε οι διαπραγματεύσει. Εμείς, ως Επιτροπή Πολιτισμού, δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουν για σας. Η Κομισιόν είναι αυτή ε, ο δικός μας που θα αποφασίσει. Ο δικός μας ρόλος είναι να είναι ασαφή η δική μας ε, θέληση. Θέλουμε να υπάρξουν πολιτιστικές ανταλλαγές και όλα όσα κάνετε, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε εξ ονόματό σα, για να μην υπάρχουν παρανοήσει. Θέλουμε να αυξηθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό για, τον, πολιτισμό, θέλουμε να προωθηθούν νέε δυνατότητε μέσω του πολιτισμού, αλλά για να είμαστε ε, ξεκάθαροι στο τι κάνει το Κοινοβούλιο και τι κάνουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ε, πρέπει να κλείσουμε όμως γιατί έχουμε και συντονιστές. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Κρίμα που η Κομισιόν δεν είπε κάτι για, την, ε, για το θέμα αυτό. Και σε σχέση με αυτά που είπε η Πρόεδρος, εγώ θα ήθελα έστω μια δέσμευση από την Κομισιόν ότι θα μιλήσετε στην, ε, στους συναδέλφους σας της Γενικής Διεύθυνσης Home και θα τους αναφέρετε το θέμα. Συνδυάστε τι εργασίε που κάνετε. Θέλουμε να προωθήσετε το θέμα των θεωρήσεων για του ε, ε, για τους καλλιτέχνες. Ε, μιλήστε και με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, μιλήστε και με την Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ. Είναι γενικές διευθύνσεις που, που πρέπει να εμπλακούν σε αυτό και θα ήθελα να το κάνετε. Ίσως όχι σε τούτη την Επιτροπή, από τη ΛΥΜΠΕ θέλουμε να προκύψει και μία πρόταση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους καλλιτέχνες. Ε, βεβαίως ε, έχουμε ε, δραστηριοποιηθεί εμείς και με τους συναδέλφους μας ε, σε αυτό που ζητάτε. Οπότε ήδη γίνεται δουλειά επ' αυτού. Γνωρίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει και γνωρίζουμε ότι και η διαδικασία για να αλλάξουν τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκη. Έχουμε ενημερώσει λοιπόν και τους συναδέλφους μας σε άλλες υπηρεσίες. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις από αυτού. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, είναι και μακροσκελής, αλλά εν πάση περιπτώσει το γνωρίζουν. Ε, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Σας διαβεβαιώ, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτά που μας είπατε. Μας ενδιαφέρει πολύ και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από αυτού. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε την συνεδρία εδώ για να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο. Οπότε όποιοι δεν είναι μέλη της, ε, των, ε, της Επιτροπής της Ομάδας των Συντονιστών παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα.